Bon, Συναδέλφοι, σα ζητώ να καθίσετε. Το 15 λεπτό των Βρυξελών έχει πλέον ήδη τελειώσει. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγή στη μερίσια διάταξη, γίνεται δεκτή. <coughs> να σας ε, μεταφέρω τις αποφάσεις τις οποίες έλαβαν χθε οι συντονιστές μας. Καταρχάς ξεκινήσαμε σε συγκεκριμένους ορισμούς εισηγητών για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού του συνδεόμενου με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού είναι η λεγόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, ε, είπαμε για τις τροπολογίες για τη διοργανική συμφωνία ανάμεσα στα τρία μεγάλα όργανα, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη δημοσιονομική συνεργασία, για μια υποδειγματική ε, δημοσιονομική διαχείριση, για την διαπραγμάτευση του κατοπήγοντος περιθωρίου και συνεισηγητές θα είναι η κυρία Τομά και ο κύριος Σόλμπρεχτ για τους δημοσιονομικούς κανόνες τους εφαρμοστέους στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα εφαρμόσουμε το άρθρο 55 για μια μεικτή επιτροπή ανάμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και τη δική μας. Και θα πρέπει να ορίσουμε ένα εισηγητή <clears throat> για την παράταση ε, δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις και για την δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου το με βάση το 55 παρατείνουμε αυτό το οποίο είχε προταθεί στα πλαίσια της, ε, του ΕΦΣΗ Euh, και ο κύριος Φερνάντες θα είναι εισηγητής. Τώρα για την αηφόρο ανάπτυξη και για την δημιουργία ταμείου εγγύσεως. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ζητά την πρώτη αρμοδιότητα και ο εισηγητής θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το Ταμείο Εγγυήσεων για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ζημίες που θα μπορούσαν να προέλθουν από την χρηματοδότηση προγραμμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι η συγγήτρια η κυρία Γκουαρδιαζάμπαλ για το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις θα είναι η συγγητής εκπρόσωπος των σοσιαλιστών για, τις, ε, ε, για τα ψηφίσματα γνωμοδότησης, για τη συνδεσιμότητα από μεμακρυσμένων τοπικών κοινοτήτων. Ο εισηγητής θα οριστεί από την ΚΟΕ. Εφαρμοστική έκθεση για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι συντονιστές ενέκριναν επίσης το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μας για το 17 αποφάσισαν οι συντονιστές για τις ακόλουθες αποστολές το 17. Την Ισία στην Πράσινη Εβδομάδα 20 με 24 Φεβρουαρίου. Παλαιστίνη ανάμεσα στις 22 με 26 Μαΐου και Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας 17ης και 21ης Ιουλίου. Βλέπετε ότι οι συντονιστές έλαβαν υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία. Αποφασίστηκαν επίσης οι εξής ακροάσεις για το 2017. Πρώτον, προετοιμασία του πολιετούς δημοσιονομικού πέραν του 2020. Υπεύθυνο γι' αυτό θα είναι ο κύριος Όλμπριχτ αλλά και η κυρία Τομά. Πέραν αυτού, χρηματοδότηση μέσω των διαφθρωτικών και επενδυτικών ευρωπαϊκών ταμείων και η σχέση των ταμείων αυτών, ο σύνδεσμός τους με άλλα ταμεία, υπεύθυνος θα είναι ο κύριος Φερνάντες. Η Έντερ Γκουαρδιαζαμπάλ για την επόμενη πρόταση για ακρόαση και επίσης ζητήσαμε να ζητηθεί εμπειρογνωμοσύνη για τις συνέργειες ανάμεσα στην συνεισφορά του κοινοτικού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών προς επίτευξη των στόχων της ετήσιας αναπτυξιακής έκθεσης. Θα είμαι εγώ υπεύθυνο. Ένα workshop για τις δημοσιονομικές πλευρές της κοινή αγροτικής πολιτικής υπεύθυνο ο κύριος Ashworth και ο κύριος Άλλη περαιτέρω ανείχνευση ε, κριτηρίων για την διαφοροποίηση προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με μειοψηφικά σχήματα. και μέσω δανείων για ε, συγκεκριμένους τομείς. Και εδώ υπεύθυνη η κυρία Γουαρδιαζάμπαλ. Υπό το φως τη συνεχούς αύξηση των ταμείων, των επιτούτου ταμείων, γύρω από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε μία μελέτη για τις επιπτώσεις αυτών των ταμείων για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Εξετάζοντας και το EFSM, και προσπαθώντας να ανοιχνεύσουμε τους κινδύνους τους οποίους εκτίθεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από τα παράλληλα ταμεία και οι επιπτώσεις των ταμείων αυτών σε χαρακτηριστικά όπως η ενότητα, η διαφάνεια και ο ετήσιος χαρακτήρας. Υπεύθυνο ο κύριος Φερνάντες. Επίσης ορίστηκε ο κύριος Νεγκρέσκου, εκπρόσωπος της Επιτροπής μας, ε, στο δίκτυο αναφορών και η κυρία Γκέριγκερ Όλτεμπεργκ σαν αναπληρώτρια. Και τέλος, σχετικά με την αμοιβή που προβλέπεται στα πλαίσια της ε, ανανέωσης ε, του απεστα, της του απεσταλμένου για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, μας από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Δράσης, δεν θα ζητηθεί με βάση το 2.23 ανταλλαγή απόψεων σε, ε, στις άλλες υπηρεσίες τις εξωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι αποφάσεις τις οποίες πήραμε χθε το απόγευμα. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις πέραν αυτών. Λάβατε όλοι επίσης μια ανακοίνωση των πρακτικών των σχεδίων πρακτικών μάλλον, των συνεδριάσεων της 24ης Ιουνίου, 14ης Σεπτεμβρίου και 15ης Σεπτεμβρίου. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συνεπώς τα πρακτικά αυτά γίνονται δεκτά. Και φτάνουμε τώρα σε ένα θέμα κρίσιμο θα έλεγα την α, αναθεώρηση ή την τροποποίηση του πολιετούς δημοσιονομικού και την τροποποίηση των οικονομικών κανονισμών. Η συζήτηση που έγινε και χθε το απόγευμα στους συντονιστές έδειξε ότι κάποια στιγμή ε, δεν θα μπορούσε να μας συνοδεύσει η κυρία Γεωργίευα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Υποτιμήσαμε την ισχύ της πορτογαλικής διπλωματικής μηχανής και η κυρία Γεωργίευα επανέρχεται euh, από τη μία είμαστε βαθύτατα θλιμμένοι γιατί πιστεύαμε ότι η κυρία Γεωργίευα είχε όλα τα χαρακτηριστικά που θα την καθιστούσαν ιδανικό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Από την άλλη εδώ και δύο χρόνια έχουμε ε, καταλήξει στο ότι έχει προσφέρει τα μάλα και ότι θα έχουμε μια ιδιαίτερο φόρο συνεργασία μαζί της και πράγματι επανέρχεται η κυρία Γεωργίεβα. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, συνεισηγητές μας, τον κύριο Όλμπριχτ και την κυρία Τομά. Ο κύριος Άλμπριχτ είναι ο πρώτος ο οποίος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για τη δυναμική αυτή διαδικασία σχετικά με την αναθεώρηση την ενδιάμεση του πολιετούς δημοσιονομικού. Υπενθυμίζω στον κανονισμό για το ΠΔΠ Υφίστερα υποχρέωση για ποσή ενδιάμεσης έκθεσης τη electoral ονομάζεται και μετά από αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση εάν κριθεί αναγκαίο, κατά περίπτωση, θα γίνει και τροποποίηση. Εμείς ως Κοινοβούλιο προτείναμε τον Ιούλιο μετά από σειρά συναντήσεων, συσκέψεων, ακροάσεων, αναλύσεων ε, υποβάλαμε την πολιτική θέση του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι βάσει των γνωσεών μας, της αναλυσής μας απαιτείται αναθεώρηση. Αυτό λοιπόν το εάν απαιτείται ισχύει. Απαιτείται. Προτείνουμε συναφώς σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά τα ανώτατα όρια, την ευελιξία και των κοινωνικούς μηχανισμούς όπως ε, όσον αφορά τις δεσμεύσεις και τις προτάσεις για την περίοδο μετά το 2020. Η Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι η προθεσμία για την έκδοση της θέσης της Κομισιόν είναι το Δεκέμβριο του 2016. Όμως η Κομισιόν ήδη υπέβαλε προτάσεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, από τον Σεπτέμβριο του 2016. Ελπίζουμε ότι η απόφαση του ΠΔΠ, η απόφαση δηλαδή, της Κομισιόν και η επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω συνένεση ε, ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εντό του 2016. Στην πρόταση τη Κομισιόν τώρα ε, υπάρχουν διάφορα στοιχεία, όπω γνωρίζετε. Το πρώτον, έχουμε τροποποιήσει για τον προπολισμό του 2017, τροποποιήσει του ΠΔΠ, του του δημοσιονομικού πλαισίου και σε 15 κυρίω χρηματοοικονομικού κανονισμού. Κύριε Τωμάκη, εγώ, οι συγητέ, οι Προτείνουμε μια κατεπίγουσα διαδικασία για να συνεισφέρουμε με τη δική μας αντίδραση όσον αφορά τις θέσεις της Κομισιόν. Η δική μας αντίδραση πρέπει να είναι ταχύτατη, σαφέστατη και τότε διότι αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε εντός του Δεκεμβρίου ο μόνος χρόνος διαθέσιμος είναι η Ολομέλεια του Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα δεύτερη του Οκτωβρίου. Προτείνουμε λοιπόν ψήφισμα, δεύτερο ψήφισμα, ε, σε ανταπόκριση της πρότασης της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή ε, ως σχέδιο τουλάχιστον θα είναι έτοιμη αύριο. Σήμερα όμως, κύριε Δωμά και εγώ, θα σα παρουσιάσουμε κάποια βασικά στοιχεία της προτινόμενης θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο εν λόγω σχέδιο επιστρέφουμε στην αρχή μας πρόταση και θυμίζουμε την πρότασή μας του Ιουλίου σε διάφορα μάλιστα σημεία του κειμένου θυμίζουμε ποια ήταν η θέση μας και ποια είναι αντίστοιχα η θέση της Κομισιόν και συνεφώς ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όπου είναι διαφορετική. Το Συμβούλιο είναι στη θέση να συμφωνήσει για την αναθεώρηση. Έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με συνένεση. Εκτός αν πούμε όχι, εμείς ως Κοινοβούλιο, στην οποία περίπτωση εμείς θα απουσιάζουμε ολοσχερό από την διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν, ως συνεισηγητές, προτείνουμε αυτό που μπορούμε να προτείνουμε, εμείς στο κοινοβουλίο που έχουμε λόγο, δηλαδή στον προπολογισμό του 2017 και εκεί συνδέουμε την κατάσταση με τον προπολογισμό του 17 και εκεί περιμένουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει κάποιες σημαντικές ουσιαστικές τροποποιήσεις. Μέρος της αναθεώρησης αφορά όντως τον προπολογισμό του 17. Και αυτό θέλω να καταθέσουμε με το ψήφισμα. Να υπάρχει σαφής σύνδεση λοιπόν με το 17. Με άλλα λόγια, εάν το, κοινο... το Συμβούλιο δεν θέλει να προχωρήσει ούτε μία αναθεώρηση, ε, εμείς ε, να τους έχουμε πιέσει όσον αφορά τον προπολογισμό του 2017. Να υπενθυμίσω επίσης και να εκφράσω την ικανοποίησή μας ότι η Κομισιόν συμφώνησε να προχωρήσει αναθεώρηση. Δηλαδή αυτό προτείνει και η Κομισιόν επί της ουσίας, προτείνει αναθεώρηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίω είναι ικανοποιητικό για μας, για το Κοινοβούλιο. Όμως, την ίδια στιγμή θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας διότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά αφορά τα ανώτερα όρια δεν ελήφθησαν υπόψη. Εμεί είχαμε προτείνει τον Ιούλιο, αν θυμάστε, ότι πρέπει να αλλάξουν τα ανώτερα όρια στον Α και στον Β κυρίω και μετά και στο 3 και στο 4. Είχαμε πει, είχαμε υποστηρίξει ότι τα ανώτερα όρια δεν επαρκούν για να πετύχουμε τους στόχους μας εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν πολιτικούς στόχους, δεν έχουμε όμως αρκετά κονδύλια. Αυτό πρέπει να το πούμε και να σωματωθεί αυτό στην αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων, των οροφών. Συναφώς να υπενθυμίσω ότι για το Horizon 2020 ε, και το Συνδέοντας στην Ευρώπη, στο μηχανισμό και στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είχαν γίνει περικοπές. Εμείς περιμέναμε, εκτιμούσαμε ότι θα ήταν διαφορετική η στάση δηλαδή ότι οι πιστώσεις θα ήταν στα ίδια επίπεδα με το 14 και το 15. Περιμέναμε λοιπόν ουσιαστική αύξηση επίσης των πόρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, το 3 και το 4. Πέρα λοιπόν των προτάσεων που είχαμε υποβάλει, και θα τα πούμε αυτά μετά και εδώ αργότερα, θέλουμε να δηλώσουμε, παραλαμβάνω, ότι είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι γίνεται θεώρηση, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα επίπεδα των πιστώσεων. Θέλω να τονίσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για την ικανοποίηση των αναγκών. Και δι, όσον αφορά τι επιπτώσει στο Horizon 2020 και στο Connecting Europe. Και δίνω το λόγο στο σημείο αυτό, στην κυρία Τωμά, για να σα πει λίγο περισσότερα πράγματα για το τι περιλαμβάνουμε στο σχέδιο αυτό ψήφισματο. Ευχαριστώ κύριε Τομά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπω είπε ο κύριο Άλμπριχτ, το θέμα είναι, το, το ψήφισμα είναι κατεπήγον, υποχρεωτικά πάρα πολύ συνοπτικό. Ε, εμείς θέλουμε όμως να είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό και γι' αυτό στην ουσία αντιπαραθέτουμε από τη μία τις προτάσεις του Κοινοβουλίου με τις προτάσεις που έκανε παλαιότερα η Επιτροπή. Και πάνω σε πολλά σημεία είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά και ε, σε κάποια άλλα οι απαιτήσει μας παραμένουν για τα μέσα ευελιξίας υπενθυμίζουμε ένα παλαιό αίτημα του Κοινοβουλίου που λέει ότι τα ειδικά μέσα θα πρέπει να υπολογίζονται μεν εκτός ανωτά του ορίου, διότι αν είχαν συμπεριληφθεί κάτω από το όριο θα επιβαρύναμε την κρίση που έχουμε στον τομέα των πληρωμών. Συνεπώς λοιπόν οι πληρωμές δεν θα μπορούσαν να γίνουν εφόσον οι πιστώσεις για τα ειδικά μέσα είχαν συμπεριληφθεί κάτω από το όριο. Συνεπώς λοιπόν αυτό το υπενθυμίζουμε γιατί δεν διευκρινίζεται από την Επιτροπή. Για την ευελιξία πάντα εμείς εκτιμούμε δεόντως τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Επιτροπή ιδιαίτερα για τις ε, υποχρεωτικές χρήσεις των πιστώσεων υποχρεώσεων. Εκτιμούμε επίσης βοηθητικά ότι το μέσο ευελιξίας και το κατεπήγον ε, ταμείο έχουν και για τα δύο προταθεί οι ενισχύσεις τους και η διεύρυνση της εμβέλειάς τους. Αλλά τα ποσά στα οποία καταλήγει η Επιτροπή είναι πολύ πιο κάτω από τα, ε, αυτά που είχαμε ζητήσει εμείς την πρότασή μας το 2016. που είχαμε ζητήσει ουσιαστικά το διπλωσιασμό. Τώρα, ε, D'abord, on se félicite que la réserve de crise qu'avait proposé le Parlement από τις απεντάξεις ή από τις απεμπλοκές εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιες προτάσεις αλλά δεν έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας. Εμείς λοιπόν εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι να χρησιμοποιείται πλήρως. Αυτή είναι η λογική του και η εκτέλεσή του πρέπει να είναι πληρεστάτη. Συνεπώς λοιπόν αυτές οι απεμπλοκές πιστώσεων δεν είναι παρά καπός της κατάστασης που λέει ότι δεν είναι αποτελεσματική η εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει το αποθεματικό για την κρίση να συνίσταται μόνο από αυτές τις, από αυτές τις αποαμπλεκόμενες πιστώσεις γιατί αν πραγματικά χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον προϋπολογισμό δεν θα έχει μείνει δίφραγκο για το Ταμείο της Κρίσης. Είναι λίγο παράλογο. Χαιρετίζουμε επίσης και την πρόταση απλούστευσης του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπως λέγεται και στην έκθεση πρωτοβουλίας, εμείς παρατηρήσαμε ότι στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου υπήρχε μια αργή ταχύτητα εκκίνησης ή και μία μη χρήση των διαφθρωτικών ταμείων, κάτι το οποίο έφτανε σε υψηλά ποσά και δημιουργούσε πολλά προβλήματα δημοσιονομικά. Συνεπώς το θέμα της απλούστευσης των κανονισμών είναι βασικό. Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει φυσικά και την πρόταση διεύρυνσης του Ταμείου Εγγυήσεων για τις επενδύσεις. Δεν πρόκειται να μπούμε στις λεπτομέρειες αυτού του νέου Ταμείου Εγγυήσεων το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξουν και άλλες εκθέσεις πάνω σε αυτό. Όμως, αυτό το οποίο θέλουμε, αυτό το οποίο ζητάμε, είναι να διευκρινιστεί πλήρως ποιες θα είναι οι οικονομικές, οι δημοσιονομικές συνέπειες αυτού του Ταμείου Εγγύησεων και ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό και η εισηγήτρια για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου και για τον προϋπολογισμό λοιπόν του 17 και για το ε, νέο πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινιστεί ακριβώς το τι αναζητούμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Τελειώνοντας το ψήφισμα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται την προετοιμασία του πολιετούς δημοσιονομικού πέραν του 20. Το είπαμε και στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας και εμένουμε ότι ε, με βάση τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει το Συμβούλιο στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Θα υπάρξουν αντίστοιχες τέτοιες αναλήψεις και για την περίοδο πέραν του 20 και για μετά το 20 και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, πρώτον για τη διάρκεια του νέου πλαισίου, να μιλήσουμε για τον επικίνδυνο, την επικίνδυνη τάση εξωτε, εξωτερήκευσης κάποιων οικονομικών μέσων πέραν του προϋπολογισμού. Και φυσικά και οι ίδιοι πόροι που είναι η βασική προϋπόθεση για έναν πραγματικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Αύριο έτσι και αλλιώ περιμένουμε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ακρόασης ε, της πρότασής σας, η οποία θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί. θα υπάρξει ψηφοφορία την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο για μια ακόμη φορά. Μου λέγουν εδώ ότι στις 12 και 10 ότι αύριο διορθώνει ο Πρόεδρος στις 12 Οκτωβρίου, όχι στις 12 και 10, θα δημοσιευθεί το σχέδιο, το σχέδιο αύριο. Και η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται την 14η Οκτωβρίου 12η Μεσημβρινή. Στις 24 πάμε πάλι στο Στρασβούργο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα κληθεί να ψηφίσει το σχέδιο ψηφίσματος. Θα υποβληθεί όπως είπα στην κρίση της Ολομέλειας την 26η και 27η Οκτωβρίου. Τώρα για τις ενδείξεις τις οποίες ε, μας μετέφεραν, τους προσανατολισμούς που μας μετέφεραν οι δύο εισηγητές, ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την πολύ και σκληρή δουλειά που έκαναν. Ευχαριστώ επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σημαντικά πράγματα που συνεισέφεραν. Η πρόταση αποτελεί μια καλή αφετηρία για την διαπραγμάτευση των θέσεων του Κοινοβουλίου. Η πρόταση όμως δεν είναι κατά βάση ικανοποιητική για μας. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για συμβιβασμό. Η αφετηρία είναι σαφής. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε αυτή την αναθεώρηση. Αλλά η αναθεώρηση καθίσταται αναγκαία, όχι επειδή τη ζητεί το Κοινοβούλιο, καθίσταται αναγκαία διότι θέλουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να αποδώσει, να λειτουργήσει και να αποδώσει, να τηρήσει δηλαδή τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Συμβούλιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επενδύσεις και άρα χρηματοδότηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται απλούστευση των κανόνων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε βελτιωμένη χρήση των ταμείων και ιδίως μέσω του διορθωτικού προηγούμενου παριθμών 4 φέτος. δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που θα θέλαμε τα επενδυτικά ταμεία και τα διορθωτικά ταμεία. Και στην ουσία βοηθούμε και το Συμβουλίο να μην χάσει την αξιοπιστία του απέναντι στους πολίτες διότι αναλαμβάνει δεσμεύσει, δίνει υποσχέσει στου Ευρωπαίου πολίτε και το μόνο που ζητούμε εμεί είναι το Συμβούλιο τελικώ να τηρήσει τα υπεσχημένα. Αυτό ζητούμε. Δεν θέλω να καταλήξω σε διαφορετικά συμπεράσματα. Θεωρώ το Συμβούλιο θα πει ναι, έχω δεσμευτεί και εκτελώ τις δεσμεύσει αυτέ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε το πλαίσιο του 2014 έως 20, το οποίο είναι μικρότερο από ό,τι για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Λέμε ότι ορισμένα πράγματα τα έχουν υποσχεθεί. Δεν νομίζουμε ότι οι υποσχέσεις που έγιναν προς επιχειρήσεις, προς πανεπιστήμια, προς τους νέους, προς τους αγρότες, προς τις περιφέρειες, και προς ποικίλους άλλους θεσμούς ότι όλα αυτά είναι νεκρογράμμα. Δεν μπορούμε να τους ε, ε, προδώσουμε όλους αυτούς. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να λένε οι ίδιες οι χώρες μέλη στους καιρούς που ζούμε. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του ίδιου φιλόδοξες όπως και το Κοινοβούλιο. Άρα το μήνυμα που δίνουμε εμείς είναι απλό. αυτά που έχουν εγκριθεί για το 2014-2020 πρέπει και να εφαρμοστούν. Αυτό είναι όλο. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζεται κάποια ευκαμψία, κάποια ευελιξία. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε τα ίδια τα ποσά των κονδυλίων, διότι το ίδιο το Συμβούλιο πρότεινε ε, να προωθηθεί η πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων. 6 δισεκατομμύρια είχαν προγραμματιστεί. Είπαν λοιπόν ότι θέλουν... Ε, Θέλω και όμως αυτό, ε, το ίδιο το Συμβούλιο τα είπε αυτά τα πράγματα. Είπε ότι τα ποσά που διαθέτουμε για την πρωτοβουλία υπέρ των νέων, υπέρ της απασχόλησης των νέων για το 2014-2020 δεν επαρκούν. Καλώς. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό. Αυτό που θέλουμε και εμείς δηλαδή και αυτό θέλει και το Συμβούλιο. Εμείς λέμε στο Συμβούλιο, ειδού οι δηλώσεις που έχετε κάνει και επιτέλους πρέπει να αναλάβετε δράση. Δράση που να δίνει αυτά αποτελέσματα. Και θυμίζω και την ε, διακήρυξη του Μακαρίδη του Σουμάν, ότι αλληλεγγύη σημαίνει ανάληψη δράσης. Με εμπνέουν τα λόγια αυτά. Οι δηλώσεις, οι διακηρύξεις του Συμβουλίου θα πρέπει να οδηγήσουν σε ανάληψη δράσης, άρα δηλαδή χρηματοδότηση, άρα χρήματα. Είμαι πεπισμένος ότι το Συμβούλιο θα πιστεί τελικώς. Επαναλαμβάνω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια ορθή βάση, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Μάλιστα, πολύ ε, φιλόδοξες οι δηλώσεις ε, Ωραία μέρα αρχίζει. Βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο που προσφέρεται για κάποια ευφορία. Εσείς τώρα κύριε Μαραγκάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Έχοντας ακούσει αυτά που είπε ο κύριος Φερνάντες, είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Η φόια λε στα γαλλικά. Πάμε. Ας δούμε λοιπόν πού βρίσκονται τα πράγματα. Αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Τομά digamos, añadir Νομίζω ότι στα πλαίσια της πρότασης για την αναθεώρηση ε, έχουν ακουστεί θα έλεγα σωστά πράγματα, υπάρχει μια λογική σειρά βλέπουμε ποια είναι τα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου Βλέπουμε το πώς θα κλείσουμε το 2016 και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια που πρέπει για το 2017. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να μείνουμε στα πλαίσια της απλής δημοσιονομικής διαδικασίας. Υπάρχει βέβαια κάποιος κίνδυνος εδώ, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βάλουμε, αν προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πάντα μέσα στο ίδιο κουτί. Αν σαν κοινοβούλιο επικρατήσουμε στις απόψεις μας αυτό θα είναι καλό. Αλλιώς όμως κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση πολύ κατώτερη από τις αρχικές μας προσδοκίες. Νομίζω λοιπόν ότι ε, σκεφτούμε ότι είμαστε τον Ιούλιο, δεν είμαστε τον Οκτώβριο. Μην τα βλέπετε τα πράγματα έτσι σε επίπεδο χρονισμού. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον τις πολιτικές ομάδες που θέλουν τα πράγματα να εξελίσσονται ορθά. Έχει προχωρήσει λοιπόν σε προτάσεις αναθεώρησης η Επιτροπή, όπως είπε και ο κύριος Φερνάνδες, δεν είναι αυτή την οποία απαιτεί και χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η ίδια η Ευρώπη απαιτεί και χρειάζεται. Και ακριβώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2013 όταν είχαμε αποδεχθεί το 14-20 το δημοσιονομικό σε επίπεδο συνένεσης και συμβιβασμού. Δεν είχαμε μιλήσει για μια βασική ριζική αλλαγή, για μια μεγάλη νίκη. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πάλι τι γίνεται με την πρόταση που είχαμε κάνει το μήνα Ιούλιο. Συμμερίζομαι και με τις παρατηρήσεις ε, και με τον κύριο Όλμπριχτ για το 1α, 1β, 3 και 4 και για τα εξωτερικά της Ευρώπης ε, οικονομικά μέσα. Νομίζω ότι σε πολλούς τομείς δεν φέρουμε εις πέρα στις υποχρεώσεις μας. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να εμείνουμε στον στόχο αύξησης σημαντικής όλων αυτών των κεφαλαίων και για την, για, το, για την Ατζέντα 2020, για το κόσμο, για το Εράσμους και τα λοιπά έχουν υπάρξει κάποιες αυξήσεις, οι οποίες όμως είναι πολύ σκαλοπιστικές οι αυξήσεις αυτές και δεν είναι ιδιαιτέρως, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία είχαμε εμείς αποφασίσει. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι η εκκρεμότητα παραμένει. Επίσης και με αυτά τα οποία ακούσαμε για το περιθώριο, το αποθεματικό για κατεπήγοντα θέματα κτλ. Και εκεί δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Συμφωνούμε πάντως με τη διατήρηση και την ενίσχυση του αποθεματικού για την κρίση Θέλουμε να διασφαλίσουμε την πραγματική του διαθεσιμότητα και την αύξηση ισχύω του. Επίσης θα πρέπει αυτά τα χρήματα, το ένα δις για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είναι σαφές ότι δεν είναι αρκετά τα χρήματα αυτά και ότι θα πρέπει να δούμε ότι το ΕΦΣΙ από μόνο του δεν μπορεί να αντισταθμίσει όλες αυτές τις όλες αυτές τις δυσκολίες. Και δεν θα μπορέσουμε έτσι να διασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης για όλους. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διαπραγμάτευση, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε ε, στο να αποδεχθούμε παθητικά σαν κοινοβούλιο ή προτάσεις μας να οδηγήσουν σε μια αλλαγή φιλοσοφίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και σε μια απίσχναση του, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το ερωτηματικό που τίθεται είναι ο προϋπολογισμός αυτός με αυτό το δημοσιονομικό εύρος μπορεί να συνεισφέρει για την καταπολέμηση των προβλημάτων μπορεί να πετύχει τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Η απάντηση δυστυχώς δεν είναι καταφατική. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πρόκληση της απασχόλησης και τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας σε πολλές χώρες. Η απάντηση και εδώ δεν είναι καταφατική. Συνεπώς λοιπόν Βλέπουμε ότι έχουμε και το πρόβλημα της ε, κρίσης της προσφυγικής μεταναστευτικής που και αυτό δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά και δεν μπορεί και ο ρόλος της Ευρώπης ε, στις ειρηνευτικές διαδικασίες πέρα των συνόρων της να ενισχυθεί και αυτός όσο θα χρειαζόταν. Λοιπόν, ας εμείνουμε στον Ιούλιο. Είπαμε, είναι Ιούλιος, δεν είναι Οκτώβριος και ας προσπαθήσουμε να οπλιστούμε σωστά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ευχαριστώ. Yes. Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ τους συνεισηγητές, εξαιρετική δουλειά, η μάδα μου. ECR θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο εκβάθρων. Ε, ποιο είναι όμως το θέμα μας. Πρώτον, το θέμα είναι πως εμείς, ε, γενικότερα ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τρία θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη-μέλη, πως, θα λέω, μπορούμε να συνοηθούμε να δράσουμε από κοινού, Και δεν μιλώ τώρα για ποιοι είναι καθαροί συνεισφορεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ομολογώ ότι εκπλήσωμε όταν κάποιοι συμπεριφέρονται ως εν... είχαμε απεριόριστα κονδύλια. Το θέμα λοιπόν πώς θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτών μας. Φέτος συνέβησαν συγκλονιστικές αλλαγές, το Brexit μεταξύ άλλων. Κανείς δεν το περίμενε, ούτε εγώ προσωπικώς. Είχα <laughs> στοιχηματίσει ότι δεν θα συνέβαινε Brexit. Εν πάση περιπτώσει, οι όροι του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Οι πολίτες δεν θέλουν... Δεν, στους πολίτες δεν αρέσει αυτός ο πληθωρισμός προγραμμάτων. Ο κόσμος είναι χωρίς δουλειές, το ίδιο και οι νέοι. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Χρειαζόμαστε προγράμματα για διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, προγράμματα για την ενεργεία. Πώς θα γίνουν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός αν είναι καλύτερο να γίνουν όλα αυτά σε επίπεδο κράτους μέλους. να το ζητήσουν, αν είναι. Μετά έχουμε ένα σωρά άλλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ας τα λύσουμε. Με, μπορούμε να τα λύσουμε με κοινού κανόνες. Πολλές φορές αυτό δεν είναι δυνατόν. Αποδεικνύεται τουλάχιστον ότι δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Συγκεντρώνουμε τις προσπαθίες μας πολλές φορές, 28 κράτη-μέλη, και οι προσπάθειε δεν αποδίδουν σε ορισμένε περιπτώσεις. Χρειάζεται λοιπόν αναθεωρήσει το ΠΔΠ, αλλά ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να δούμε ποια είναι τα βασικά μας προβλήματα. Ας περιοριστούμε στα βασικά, τα ουσιαστικά προβλήματα και ας συγκεντρώσουμε τα μέσα που διαθέτουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε επιπλέον κονδύλια για κάποιες επιμέρους πτυχές των προβλημάτων, σύμφωνοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τα κρατημέλη, άρα λοιπόν αυτό το περιμένουν τα κρατημέλη, τα, οι πολίτες μας, με συγχωρείτε από εμάς. Οπότε το να λέμε απλώς ότι θέλουμε περισσότερες πιστώσει δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ. Το θέμα είναι να συγκεντρωθούμε στα ουσιαστικά. Λοιπόν, η πεπατημένη δεν θα μας βγάλει πουθενά. Ναι, λοιπόν, στην αναθεώρηση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, αλλά ποιοι είναι οι στόχοι, ποιε είναι οι προτεραιότητε. Να αρχίσουμε προτεραιότητε για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια. Να αναρωτηθούμε, οι προτεραιότητε του χθε ισχύουν σήμερα. Ας ε, πάρουμε τη Γεωργία, για παράδειγμα. Δεν είναι κινδυνεύμα να πεινάσει κανείς πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η μετανάστευση είναι μια νέα πρόκληση. Πώς εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ κύριε Γκέσλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οποία μας είπε η, κυρία Τομά και ο κύριος Σόλμπριχτ παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε επίπεδο ελέγχου προϋπολογισμού είναι επίγον να υπάρξει μια πιο αξιόπιστη εικόνα ε, σε σχέση με τα μέσα αυτά. Τα μέσα τα οποία βρίσκονται εκτός του τακτικού προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμεύουν στην βελτίωση των ισογισμών των πιστοτικών ιδρυμάτων, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος και θα πρέπει το, η προβληματική αυτή να εμβαθυνθεί περισσότερο. Αυτό που λέει η κυρία Τομά, ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία στην παρούσα φάση σκιάζονται από άλλα και θα πρέπει να τα φέρουμε στην επικαιρότητα θα πρέπει να μην βέβαια απαιτούμε όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τόσο το καλύτερο. Οι δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν δεν είναι δράσεις τις οποίες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι δράσεις που ανήκουν σε κάθε μία ε, κυβέρνηση κράτου μέλους. Τώρα το θέμα που τίθεται είναι γιατί δεν έχουμε τις αρμοδιότητες αυτές, ε, γιατί δεν έχουμε τη νομική βάση και είμαστε υποχρεωμένοι να ξοδευόμαστε σε αναποτελεσματικές παρεμβάσεις. Ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες αποτυγχάνουν διότι δεν εκτελούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Έχω και κάτι ακόμα για το MFF, το ερώτημα δηλαδή του Brexit. Γνωρίζουμε τώρα ότι οι Βρετανοί βεβαίως δεν έχουν υποβάλει ακόμα την αίτηση, αλλά το θέμα αρχή είναι τι κάνουμε με την κοινή περιουσία και με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αποχωρεί ένα μέλος. Βασικό θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Πρώτο ερώτημα λοιπόν. Τι κάνουμε στην περίπτωση που αποχωρεί μια χώρα μέλος και επομένως προκαλείται ένα κενό. Θεωρητικό ερώτημα, αλλά πρέπει να συζητηθεί. Και δεύτερο, τι κάνουμε με το συνότυπο σου έχουμε 8,7 δισεκατομμύρια ε, ε, περιουσία, αλλά υπάρχει όμως και περισσότερο ε, ύψος χρεών. Δηλαδή τελικώς το υπόλοιπο είναι αρνητικό. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και θα βοηθήσουν πολύ και στις περαιτέρω συζητήσεις. Κοιτάξτε, κύριε το Brexit μπαίνει στη ζήτηση των πραγμάτων. Θα επηρεάσει το δεύτερο μέρος του ΠΔΠ. Σύμφωνοι υπάρχουν κάποιες ε, αβεβαιότητες που θα προκύψουν 18, 19, κάπου εκεί. Ούτως ή άλλως ο Χωσέ Μανουέλ θα μιλήσει για το θέμα. Κάποιες απολύσεις θα έχουμε σίγουρα, λόγω Brexit. Οι πρώτες ε, αφορούν την ισοτιμία της λίρας με το ευρώ και θα χάσουμε κανένα δισεκατομμύριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι προηγούμενοι είπαν περισσότερα από αυτά τα οποία θα είχα να πω. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο γενικά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία είναι καλή πρόταση γιατί ακολουθεί πολύ στη γραμμή την οποία θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσουμε για τα μέσα ευελιξίας τα οποία ορίζουν αν θέλετε το ευρύτερο πλαίσιο και για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές ορίζουν επίσης και την τροφοδοσία ε, του αποθεματικού για την κρίση όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά στην ουσία γίνεται με απεμπλοκές πιστώσεων ε, οι αποδεσμεύσεις πιστώσεων για να έχουν δηλαδή χρήματα διαθέσιμα τα ταμεία αυτά και ιδιαίτερα το αποθεματικό για την κρίση θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται με ικανοποιητικό τρόπο στον προϋπολογισμό. Πάντως το θέμα της ευελιξίας πάει καλά από πλευρά των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα σε επίπεδο αριθμών βέβαια η κατάσταση δεν είναι ποσοτικά εννοώ ε, ικανοποιητική. Ε, για το σχέδιο Juncker σαν παράδειγμα χάνει το πρόγραμμα ε, Ευρώπη, μάλλον Ατζέντα 2020 τουλάχιστον 400 εκατομμύρια. Συνεπώς λοιπόν είμαστε πολύ μακριά από αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν περισσότερα χρήματα γιατί κατά τα άλλα δουλεύουν καλά τα προγράμματα αυτά όπως το Erasmus Plus και το COSME. Τώρα για την εγγύηση για την απασχόληση των νέων και θα απαντήσω και στην κυρία Γκρέσλε γιατί εδώ διαφωνώ μαζί της. Είναι προφανές ότι η απασχόληση των νέων δεν είναι ένας χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων ή όχι, μπορεί να είναι συζητήσιμο. Αν η απασχόληση γενικά είναι εθνικό θέμα. Αλλά η αλληλεγγύη είναι ευρωπαϊκό θέμα. Και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προφανώς υπεύθυνη για όλες τις χώρες και τις πλούσιες και τις φτωχότερες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε τα ταμεία με στόχο την αλληλεγγύη και ακριβώς γι' αυτό δημιουργήθηκε το ταμείο αυτό και θα πρέπει να είναι λειτουργικό. Γιατί σε ορισμένε χώρες τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα. Δεν είναι θέμα χωρών, είναι θέμα κοινωνικό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ ψηλή και θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί καλύτερα η πρωτοβουλία για τους νέους Είδαμε ότι η αξιολόγηση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα είναι μια θετική, αλλά υπάρχει σαφώ χώρο για βελτιώσεις γιατί να καλυφθούν οι ανάγκε. Και ένα γενικότερο σχόλιο τώρα, το οποίο ε, θα ήθελα να σταλεί σαν μήνυμα στο Συμβούλιο. Δυστυχώ, η εμπειρία μέχρι τώρα μα δίδει δίκαιο, μα δικαιώνει. Κάθε φορά που λέμε εμείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, σημειώνουμε το πρόβλημα. Κάθε φορά που λέμε ότι υπάρχει μια ανάγκη, ότι υπάρχει μια προτεραιότητα ή μια έλλειψη χρηματοδότησης, τότε πραγματικά δεν έχει νόημα να επιμένει κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το είδαμε επίσης και με την ευελιξία όταν διαπραγματευθήκαμε το δημοσιονομικό πλαίσιο και σε δυόμισο χρόνια είδαμε τον περιορισμένο περιθώριο ευελιξίας του προϋπολογισμού είδαμε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες για τους στόχους ε, που έθεσε και που ανέφερε και ο κύριος Μαραγκάη και είμαστε πολύ μακρά, αλλά έστω μόνο και μόνο για να έχουμε μια ευπρεπή παρουσία στους τομείς αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα κατανοήσει κάπως καλύτερα αυτά τα οποία ζητάμε και θα κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο και να μπορέσουμε ε, να δείξουμε στους συμπολίτε μας ότι τα πράγματα τα παίρνουμε σοβαρά και όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό μιλάμε για τα προβλήματα των ανθρώπων, των νέων, των προσφύγων και ότι υπάρχει δυνατότητα να διορθώσουμε αυτά τα οποία χρειάζεται στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό. Ελπίζω τα πράγματα να βελτιωθούν έστω και λίγο. Ευχαριστώ. Κύριο Στενένο πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τους δύο εισηγητές, ιδιαίτερα για το κατεπήγον ψήφισμα το οποίο πρέπει να έχει αντίκτυπο. Πρέπει να κρατήσουμε τη θέση μας σαφή. Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα Χρειαζόμαστε περισσότερη λοιπόν ευελιξία. Τώρα όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη χρηματοδότησή τους, να το δούμε. Οι προτάσεις ε, της Επιτροπής δεν είναι επαρκής για το 1α, 1β, 3 και 4 δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Δυστυχώ δεν έχουμε να κάνουμε μια ενιαία πολιτική, είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία όμω εμεί πρέπει να υποστηρίξουμε. Δείτε στι ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί στηρίζουν τη γεωργία του ε, κατά κεφαλήν δύο φορέ περισσότερο από ό,τι η Ευρώπη και οι Κινέζοι το κάνουν τρει φορέ περισσότερο από ό,τι η Ευρώπη. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Να στηρίξουμε τη γεωργία μα που, εντάξει, η γεωργία είναι ένα ειδικό τομέα, εξαρτάται από το κλίμα, από τις ανάγκες τη υγεία κλπ. Συν η πίεση από του οικολόγου. Λοιπόν, η Γεωργία, παρατορή συνάδελφο, λέει ότι κάναμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε ω Ευρώπη για την Γεωργία, για το οποίο δεν είμαι πεπισμένο, αλλά αυτό γίνεται και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει προφανώς τα πλεονάσματα ως ανθρωπιστική βοήθεια, καμία αντίρρηση. Αυτά θα τα δούμε στο κεφάλαιο 2. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Κουντή. Ευχαριστώ. Έχουμε θέματα εδώ Έχουμε και το θέμα της ισοτιμίας και το πώς θα μας επηρεάσει με την λίρα. Είναι το πρώτο το οποίο θα καταβάλει η χώρα μου. Πληρώνουμε, θα πληρώσουμε και αυτό μετά από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Πάντως θα είναι μακρά η πορεία. Να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Το άρθρο 50 δεν έχει κινητοποιηθεί, δεν έχει θερμολογηθεί. Δεν έχουν καν ξεκινήσει οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την έξοδό μας. Οπότε, συνάδελφοι, μην προτρέχετε. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε αρτήσει βεβαίω των εξελίξεων και των διαπραγματεύσεων και της εξέλιξης της σχέσης των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα το έργο της Σεμπέλα και του των δύο συγκεκριτών εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την αναθεώρηση του ΠΔΠ. Έχω μια ερώτηση. Θα το δούμε και στη συνέχεια βεβαίω. Τι είναι η το FC2 και τι επιπτώσει στον προπολογισμό. Ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του προπολογισμού αφήνονται σε επιδυτικές πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω όμως η πρώτη αναθεώρηση που θα οδηγήσει Νομίζω ότι ο προπολογισμό πάντως πρέπει να διατηρήσει τον ρόλο που έχει να είναι προπολογισμό και να μην είναι πανά σε έκτακτε πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι. Συμφωνώ με τους περισσότερους εκ των συναδέλφων μου που εξέφρασαν άποψη για το EMFF πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες, δηλαδή ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Αυτά υπάρχουν ε, σχέδια τα οποία είναι πάρα πολύ, ε, είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είπε ο κ. Γιούνκερ ότι στις αρχές του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε 2,4 εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Και χάρη στην πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την στήριξη της νεολαίας. Εμείς συμφωνούμε όλοι. Και ο κ. Γιούνκερ, γιατί άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει δέσμευση για το 2016 για να υλοποιηθεί το 2017. Ενώ αυτή είναι η πρώτη πρώτη προτεραιότητά μας. Και βλέπουμε να υπάρχει και κάποια σημαντική απόδοση, μια σημαντική επιτυχία. Εάν ρωτήσετε εκπροσώπους χωρών μελών, θα σας πούν ότι οι νέοι, όταν έχουν λάβει μια υποστήριξη για ένα εξάμεινο, για παράδειγμα, ένα υψηλό ποσοστό εξ αυτών διατηρούν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν μπορέσει να κατακτήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να διαθέσουμε κονδύλια στον προπολογισμό για την στήριξη της πρωτοβουλία αυτή, διότι αξίζει τον κόπο. Βρίσκουμε δουλειά σε ανθρώπους και πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία γιατί οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται πλέον στην αγορά εργασία και παραμένουν σε αυτήν. Εγώ είμαι απογοητευμένο, διότι ενώ το project αυτό έχει αποδείξει την επιτυχία του, δεν μπορέσαμε να το αξιολογήσουμε μέχρι το 2016. Έχουμε χάσει την πραγματικότητα, αφού έχει ξεκινήσει το 2014, δύο χρόνια. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Να μην παραμείνουμε στις θεωρίες. Χρειαζόμαστε ορθή διαχείριση γιατί αυτά τα πράγματα καρποφορούν. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και να το αποδώσουμε υψηλή προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Φτάνουμε πλέον στο τέλος της ανταλλαγής απόψεων για το σχέδιο ψηφίσματος που έχουν συντάξει οι δύο συνεισηγητές στη συνέχεια σημαντικών εργασιών για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή όταν το ΠΔΠ εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2013, το φθινόπωρο του 2013, δεν είχαμε προβλέψει την κρίση που θα προέκυπτε από την μαζική μετανάστευση και που οδήγησε βεβαίως, μάλλον που προήλθε από την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της υποσαχάριας Αφρικής. και βεβαίω με την πόρτα που άνοιξε όταν κατέρευσε το λιβικό καθεστώς. Βεβαίω δεν ε, πρέπει να ζητούμε περισσότερε δαπάνες. Αυτό που είναι ο ρόλο μα είναι να καταδείξουμε ότι όταν ζητούν οι χώρε μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει κάποια δράση για λογαριασμό τους, οι χώρε μέλη μεν εξοικονομούν, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να αποδείξουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία με τις δράσεις που αναλαμβάνει. Βεβαίω πρέπει να ευρεθούν και τα ορθά επιχειρήματα για να πιστεί το Συμβούλιο. Με το να επιμείνουμε στο μήνυμα το οποίο αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη οποιασδήποτε χώρα μέλου. Διότι εύκολα μπορεί να πει το Συμβούλιο ότι, α, κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπερβολικά γενναιόδωρο. Δεν πρέπει να πέσουμε όμω σε αυτήν την παγίδα και να εκτεθούμε σε τέτοια κριτική. Να δώσουμε δηλαδή ε, τον ρόλο του καλού στο Συμβούλιο, διότι αυτό σφίγγει τι στρόφιγγε. Πρέπει να δείξουμε ότι αυτά που γίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν κάτι δεν μπορούν να το αναλάβουν οι ίδιε οι χώρε μέλη, ότι γίνεται καλύτερα όταν αναλαμβάνει τα ενία η Ευρώπη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ε, εισηγητές μας ότι θα εύρουν τα κατάλληλα επιχειρήματα διότι πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και όχι μόνο στο Συμβούλιο. Και όταν θα το έχει κατανοήσει αυτή, αυτό η κοινή γνώμη θα ασκήσει με τη σειρά της πιέση της κυβερνήσης των χωρών μελών και το Συμβούλιο θα τίνει πλέον ευήκονους στις ε, επιθυμίες και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι και εσάς κύριε Τωμά και εσείς κύριε Όλμπριστ. Α, εσείς θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω να πω ότι πρώτα πρώτα ευχαριστώ ε, όλες και όλους τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους. Υπενθυμίζω ότι οι θέσεις μας και του Ιουλίου και η τωρινή που έχει προκύψει και από τις ακροάσεις και αναλύσεις που έχουμε κάνει. Δεν πρόκειται δηλαδή για πολιτική θέση η οποία επιζητεί την αλλαγή για χάρη της αλλαγής. Έχοντας κάνει την ανάλυση των γεγονότων διαπιστώνουμε ότι το σύστημα χρειάζεται τροποποίηση, αναθεώρηση. Διότι αν δεν γίνει αυτό όταν θα έρθει το Brexit το σύστημα δεν θα μπορέσει να αντέξει. Άρα δεν πρόκειται για βολονταριστική θέση του Κοινοβουλίου που επιθυμεί να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στα του προπολογισμού. Δεύτερο, στο ψήφισμά μας με την συζήτηση για την ορθή χρήση των κονδυλίων. Αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει και με μια σε βάθος απλούστευση των διαδικασιών και κανόνων. Δεν αρκεί απλώς να μετακινηθούν κονδύλια από μια θέση σε άλλη. Χρειάζεται και η απλούστευση, όπως είπα, που είναι στοιχείο κλειδί. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 να υπάρχει η νέα πρόταση δημοσιονομικής προοπτικής. Άρα, έχουμε γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Τώρα έχω και το εξή. Μέσα στον κανονισμό προβλέπεται η αναθεώρηση να αφορά τις προτεραιότητες. Μπορούμε να καταδείξουμε ίδιο, τόσο ότι η κατάσταση έχει αλλάξει από ότι πριν από μία τριετία. Έχουν αλλάξει λοιπόν οι προτεραιότητες. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Υπάρχει η πρόκληση των προσφύγων και βεβαίως και η Βρετανική έξοδος. Άρα χρειάζεται, χρειάζεται να γίνουν νέες επιλογές και νομίζω ότι οι θέσει των συναδέλφων μας εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ενισχύουν την θέση και την εργασία μας. Απαντώ στον κύριο Κορνέλ ότι ο μηχανισμός που υποτίθεται ότι θα μειώσει την γραφειοκρατία και ότι στην βάση αυτών μετά θα μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια. Καταρχήν είμαι σύμφωνο. αλλά μπορεί ωστόσο να περιπλακούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και ίσω να αποδειχθεί ότι είναι και υπερβολικά αργά για να ζητήσουμε νέα κονδύλια όταν θα έχει ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική απλούστευση. Πάντως είμαι σύμφωνο μαζί σα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εάν δεν βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών. Και τελευταία παρατήρηση κύριε συνάδελφε. Τον Ιούλιο προτείναμε τα κονδύλια, οι πιστώσει να παραμείνουν στο υπερβάλλουσες πιστώσεις, δηλαδή να παραμείνουν στο προπολογισμό. Τελικώ αυτό αποδεικνύεται δύσκολο και καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Στο προσχέδιο 4 έχουμε 7 δισεκατομμύρια τα οποία θα επιστραφούν στις χώρες μέλη. Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Δεν ζητούμε περισσότερα χρήματα εμείς, αλλά να παραμείνουν τα χρήματα στον προπολογισμό. Γνωρίζουμε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών θέλουν να του επιστραφούν τα κονδύλια αυτά. Το κοινό ωστόσο πρέπει να κατανοήσει με το επιχείρημα αυτό ότι εμεί δεν ζητούμε περισσότερα χρήματα αλλά, ε, ζητούμε καλύτερη διαχείριση των υφισταμένων κονδυλίων. Και ότι είχαμε δίκιο που το προτείναμε εξ αρχή. Ευχαριστώ κύριε Όλμπρεκτ για τι ευκρινήσει. Ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να προσπαθήσω να πείσω τους περισσότερους εδώ, αν και είναι ήδη πεπισμένοι ότι δεν είναι σκοπός μας να ζητήσουμε περισσότερες πιστώσεις. Και στο κάτω-κάτω για ποιον, γιατί εδώ το 99% τους άλλους των πιστώσεων επιστρέφει στα κράτη-μέλη. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Και ο Φερνάντες το είπε, εμείς θέλουμε να είμαστε απλώς ρεαλιστές καθένας από εμά ε, εμφορείται από τις δικές του εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και ευαισθησίες. Εμείς τι κάνουμε εδώ τώρα. Καταδείξαμε, πιστεύω, ε, το είπε και ο πρόεδρος νομίζω, ότι σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έρχεται το Κοινοβούλιο να ανακοινώσει ναι μέτρα, νέου μηχανισμού. Όχι, αυτά τα κάνει το Συμβούλιο. Εμεί λοιπόν, όσο πιο ρηκημερικά γίνεται, διαπιστώνουμε το χάσμα το μεταξύ πολιτικών διακηρύξεων και των μέσων τα οποία τίθεται στη διάθεσή μα για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία, για την Ευρώπη, για την πολιτική. Διότι έτσι την αξιοπιστία του οι πολιτικοί. Λόγια χωρί ε, πράξει είναι η τέλεια συνταγή για την απαξίωση της δημοκρατίας μας, για την απώλεια της εξοπιστίας μας. Συνεπώς, θα το ξαναπώ, δεν είναι ότι δεν είμαστε αρκετά Ευρωπαίοι εδώ, ότι δεν υποστηρίζουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όμως ας είμαστε ρεαλιστές. Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Χρειάζεται ένα ελάχιστο ρεαλισμού για να καθιερώσουμε και να υλοποιήσουμε αξιόπιστες πολιτικές. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμά μας. Και το λέω αυτό προς τον συνεισηγητή μου. Δεν ξέρω αν πρέπει να στείλουμε ένα ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα, γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε πάρα πολύ λογικοί νομίζω. Πολύ προσγειωμένοι και δεν θέλω να αρχίσω να κατηγορώ, αλλά για είμαστε μάρτυρες ε, απίστευτης μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από κάθε σύσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να είμαστε προσγειωμένοι και να στείλουμε το μήνυμα ότι οι γενικές πολιτικές κατευθύνσεις πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέσα. Καλές πρωτοβουλίες για την ανέργεια των νέων ή για την γεωργία. Αυτά α τα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα δεν είναι να τα συζητάμε στι επιτροπέ, στι ειδικέ επιτροπέ. Η κατεύθυνση έχει προκριθεί, έχει ψηφιστεί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση σας φροντίσει να βρει τα μέσα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε αμερόληπτα, ισορροπημένα και ως Ευρωπαίοι. Πρόεδρος, κλείνει η συζήτηση επί του θέματος. Πάντως νομίζω ότι έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι βρισκόμαστε στο τέλος ενός κύκλου όπου οι προπολισμοί δεν λειτουργούν επαρκή μέσα. Είναι θεσμικό το πρόβλημα γιατί τι είναι προπολισμό εν τέλει, είναι η έκφραση ενό πολιτικού εγχειρήματο. Πολλέ φορέ λοιπόν έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν όχι όλα, έχουν περισσότερο στο μυαλό του τι επόμενε εκλογέ και δεν μπορούν, να, δεν μπορούν να πάνε παραπέρα από τι επόμενε εκλογέ στη χώρα του. Αυτό το οποίο υπογράμμισε, το Τωμάς, είναι ότι το μεγαλύτερο χάσμα είναι μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Εγώ ασχολούμαι με τις πληρωμές γιατί αυτά εμφαίνονται στον ετήσιο προπολισμό, αλλά το χάσμα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Το είπε και ο κύριος Σόλμπριχτ όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία και τους κανόνες για τον προϋπολογισμό θέμα είναι να μιλήσουν οι θεσμοί στους πολίτες. Να μας πούν αυτοί πώς αντιλαμβάνονται την Ευρώπη. Ανταποκρίνεται η Ευρώπη στις προσδοκίες. Τι γίνεται όταν κάποιος ζητάει και μια μικρή χρηματοδότηση. Πρέπει να συμπληρώσει δεκάδες σελίδων, να αφιερώσει ατελείωτο χρόνο για να γίνει μια μικρή ενίσχυση. Το ξέρω από την έρευνα ένας ερευνητής μου έλεγε ότι υπάρχουν ειδικά γραφεία τα οποία εισπράττουν τέλος επιτυχίες, αμοιβή επιτυχίες. Αναλαμβάνουν λοιπόν να υποβάλουν αιτήσει στην Κομισιόν και λένε ότι τους ερευνητές για παράδειγμα, εάν πάρουμε τη σύμβαση, την επιδότηση, θα μου δώσετε τόσο της εκατό του προπολογισμού σας. Αυτά δεν είναι πράγματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει τα χρήματα εκεί που πρέπει και όχι στη γραφειοκρατία. Λοιπόν, να απλουστεύσουμε τους κανόνες, να βάλουμε μία τάξη. Παρός, πολλές φορές και εμείς νομοθετούμε, κάνουμε τα πράγματα πιο πολύπλοκα, θεσμοθετούμε υπερβολικά πολλούς κανόνες για εκ των προτέρων ελέγχους, και ξεχνούμε πολλές φορές την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή απορρίπτουμε ένα έργο, μια πρόταση, επειδή λείπει ένα βιογραφικό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αντί να ασχοληθούμε με την ουσία ενός έργου, μιας πρότασης, το οποίο είναι και η ουσιαστική δυσκολία. Αυτά. Θα ήταν ατελής η ανταλλαγή απόψεων εδώ αν δεν ακούγαμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επέστρεψε η κυρία Γεωργίευα. Ναι, ναι, επέστρεψε στις 24 ώρες μετά την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια χαρά, ζητά συγγνώμη, δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα. Ε, θα της πείτε ότι αντιπροσωπεύθηκε πλήρως και θα είναι παρούσα και για τον τριμερή διάλογο και για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Να μου επιτρέψετε παρακαλώ να κάνω τρία σχόλια μετά από τη συζήτηση αυτή, την οποία θεωρώ ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Πρώτον θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την προσπάθεια που κάνει. Οι συγητές του έκαναν εξαιρετική δουλειά και με χαρά άκουσα ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά είστε ικανοποιημένοι και από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίρνουμε κομπλιμέντα γι' αυτό μας χαροποιεί. Έτσι κάναμε προσπάθεια για να κάνουμε μια πρόταση φιλόδοξη αλλά και αξιόπιστη και λογική. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ότι τα στοιχεία μας είναι θετικά. Θα ήθελαν σε προσωπικό επίπεδο να προχωρήσουν πέραν αυτών αλλά Είδατε ότι τα στοιχεία που έχουμε προτείνει είναι θετικά. Δεύτερο σχόλιο. Σκοπεύουμε να καταθέσουμε μια διορθωτική επιστολή ε, για να μεταφράσουμε αν θέλετε ε, τις αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού στον επόμενο προϋπολογισμό. Και τρίτο σχόλιο. Να διευκρινίσω κάτι που είπε η κυρία Τομά ότι εμείς δεν ήμασταν ξεκάθαροι σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τα λεγόμενα ειδικά μέσα και αν είναι πάνω από το ε, όριο του πολιετούς. Εμείς διευκρινίζουμε ότι σαν Επιτροπή πάντα υποστηρίξαμε ότι οι πληρωμές αυτές είναι πέραν του ορίου και οι προβλέψεις μας για τις πληρωμές ε, μέχρι το 2020 οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις που συνόδευσαν την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού βασίζονται στην αντίληψη ότι οι πληρωμές για τα ειδικά μέσα είναι πέραν του του ορίου και γι' αυτό ακριβώς διευκρινίσαμε προς το Συμβούλιο ότι οι νομοθετικές μας προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού χωρίς να τροποποιηθούν τα όρια που είχαν γίνει δεκτά το 2013. Περιμένουμε λοιπόν την τελική πρόταση από πλευρά σας και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πριν το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ κυρία Καλβίνιο. Νομίζω ότι βασικός στόχος αυτής της διαπραγμάτευσης είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις διαφορές ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Υπήρχε συμφωνία σε σχέση με τις υποχρεώσεις για το πέραν του ορίου, αλλά όχι για τις πληρωμές. Εντελώς υποκριτική η κατάσταση και γι' αυτό ένας από τους στόχους της διαπραγμάτευσης θα είναι να αναγνωρίσει επιτέλους το Συμβούλιο ότι και οι πληρωμές είναι στην ίδια κατάσταση με τις υποχρεώσεις για τα λεγόμενα ειδικά μέσα. Λοιπόν, θέλουμε λίγη τύχη εδώ. Κοιτάξτε, αν το πούμε έτσι όπως το λέμε θα το καταλάβει και ε, η κοινή γνώμη. Αλλά όταν λέμε ότι ναι μεν οι υποχρεώσεις είναι εκτός αλλά οι πληρωμές εντός αυτό μπερδεύει τον κόσμο και δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ε, κύριε Όλμπρεχτ και κυρία Τομά περιμένουμε την τελική σας πρόταση και σας συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά. Θα περάσουμε τώρα στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Για το 2016, τον τέταρτο. Και αν ο κύριος Φερνάντες μας το επιτρέπει, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με την τέταρτη και με την πέμπτη επιστολή. Ρυθμίσεις σχετικές με την πρόσφατη επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Την πήραμε την προηγούμενη Παρασκευή. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης και το θέμα ακριβώς για τους ιδίους πόρους. Να πω ότι είχε υπάρξει και στο παρελθόν μία τροποποίηση, εδώ και δύο χρόνια μάλλον, ειδική για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε κάθε δύο χρόνια να υπάρχουν τροποποιήσεις για τους ίδιους πόρους. Πώς πάει ακριβώς η υπόθεση. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε κάπως καλύτερα. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 16. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο διορθωτικός λοιπόν υπαριθμών 4. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε σεβαστές τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει και μάλιστα σε ύψος 7 δις για την πολιτική συνοχής. 7 δις είναι λοιπόν το ποσό το οποίο είχαμε αναλάβει την υποχρέωση να καταστήσουμε διαθέσιμο και το οποίο θα καταλήξει στις τσέπες των κρατών μελών. Συνεπώς λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι υποχρεώσεις οι οποίες είχαν αναλυφθεί στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης γενικότερα των τοπικών περιφερειακών αρχών, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των επενδυτικών σχημάτων για την ευφυή ανάπτυξη. Όλα αυτά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα τιμήσουμε σε εισαγωγικά. συνολικά για τις 28 χώρες και τις εκατοντάδες περιφέρειες. Επτά δις λοιπόν ξαναγυρίζουν στις τσέπες των κρατών μελών και αυτό είναι αρνητικό για την κατάσταση αυτή. Τα χρήματα αυτά τα είχαν υποσχεθεί και ε, για τις πιστώσεις αυτές θα υπάρξει αναβολή καταβολής τους. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο επί της ουσίας, είναι και γραφειοκρατικό γιατί βρέθηκαν επτά δις που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά νομίζω τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Το Συμβούλιο είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης. Έχω την αίσθηση ότι ε, ε, η μισή από τους υπεύθυνους που είναι, θα έλεγα, στις λεγόμενες διαχειριστικές αρχές δεν έχουν ακόμα διοριστεί. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είναι απαραίτητο για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την σοβαρότητα η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον σεβασμό των ανηλυμένων αποφάσεων να υπάρξει μια αναθεώρηση ε, του πολιετούς δημοσιονομικού. Απαιτείται περισσότερη δημοκρατία, απαιτείται περισσότερη γραφειοκρατία ε, και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Ε, αναφερόμαστε σε μία μείωση λοιπόν των πιστώσεων πληρωμών κατά 7,2 δις. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα σοβαρά για τις πληρωμές στο μέλλον. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα τα οποία έχουμε ήδη ε, υποσχεθεί, είναι χρήματα τα οποία έχουν προϋπολογιστεί αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστώσεις. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο έτσι ώστε να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας και τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον στόχο για τον οποίο προβλέφθησαν. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργήσει προληπτικά σε σχέση και με ε, το ΕΦΣΥ με το στρατηγικό ταμείο. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα αποφάσεις για την παράταση του ΕΦΣΥ eh, e Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βασιζόμαστε στην αρχή η οποία λέει ότι το ποσό που θα αποφασιστεί μπορεί και να μην είναι απόλυτα απαραίτητο διότι δεν είναι σαφές ότι το 2016 θα διασφαλιστεί η παράταση ε, της ισχύω του ΕΦΣΙ στο τέλος του 16 μέχρι το τέλος του 16. Στον τίτλο 3 επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα ξεχωριστό το οποίο τίθεται λόγω των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών υπάρχουν 250 εκατομμύρια ε, υποχρεώσεων και 275 πληρωμών. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, σχετικά με τον διορθωτικό 4. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Αναφερόμαστε σε πιθανές διορθώσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για το Ηνωμένο Βασίλειο. 730 εκατομμύρια δόθηκαν επιπλέον λοιπόν το 2012. 361 για τις διορθώσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2015. Υπάρχουν όμως και άλλες ε, μορφές αντιστάθμισης ε, που δεν λάβαμε υπόψη. Σαν παράδειγμα ε, Υπάρχουν κάποιες επιστροφές προς τέσσερις χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες. Οι διορθώσεις αυτές λοιπόν δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες, δεν είναι σαφείς. Στα πλαίσια λοιπόν του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαρίθμου 4 προβλέπεται ένα δις περίπου για τα πρόστιμα και για την αντιστάθμιση των ε, τη μείωση της αξίας της στερλίνας απέναντι στο ευρώ. Και εδώ ίσως θα πει να προβλεφθεί μια αντιστάθμιση. Και τίθενται εδώ και ορισμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμούν τέσσερα λοιπόν αναφερόμαστε στην ε, ε, εκτέλεση του μύθ κατά 100%. ...100% λοιπόν για το αμύφ. Αλλά μόνο το 10% των δαπανών αυτών έχουν ήδη ξεκινήσει για τους πρόσφυγες, επαναλαμβάνω, και τις διαδικασίες επανεγκατάστασής τους. Τελικά τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν πλήρως στα πλαίσια της απόφασης για τις επανεγκαταστάσεις. Και μια άλλη ερώτηση η οποία τίθεται και αναφέρομαι τώρα για τον διορθωτικό υπαρίθμο 5 απαντώντας και στον πρόεδρό μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πανεπιστημιακό δίπλωμα για να μπορέσει κανείς να καταλάβει πραγματικά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπάρχει μια τεράστια σύγχυση ανάμεσα στους ιδίους πόρους από τη μία ε, και στις ε, τις απαλλαγές από την άλλη και τις εξαιρέσεις επί των απαλλαγών ή τις αποκλήσεις επί των απαλλαγών. Λοιπόν, απαιτείται μεγαλύτερη απλότητα σε σχέση με τους ιδίους κυρίως πόρους έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμος εισαγωγικά από όλου τους πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης ο κοινότικό προϋπολογισμός. Αυτό ισχύει και για τους Βρετανού και για τους Σουηδού και για τους ε, Ολλανδούς και για τους Αυστριακού κτλ. κτλ, κτλ. Τώρα, ε, για τους ιδίους πόρους πάντα απαιτείται μια βελτίωση από πλευράς, ε, μια αύξηση ουσιαστικά δηλαδή από πλευράς όλων των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία επιστρέφονται σημαντικά ποσά. Υπάρχουν όμως και άλλα κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν παίρνουν τα χρήματα που θα ανέμενε κανείς. Συνεπώς λοιπόν εμείς ε, έχουμε μία συγκεκριμένη άποψη σαν κοινοβούλιο σε σχέση με τις εθνικές συνεισφορές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο καθορίζονται αλλά και με ποιο τρόπο εκτελούνται οι συνεισφορές των κρατών μελών έχουν προβλεφθεί σαν παράδειγμα για την δημοσιονομική περίοδο 2017. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τον διορθωτικό υπαριθμόν 5 για να λάβουμε υπόψη μας τις προσδοκίες των κρατών μελών να γνωρίζουν τι θα τους περιμένει στα πλαίσια του επόμενου προϋπολογισμού. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστούν καλύτερα τα πράγματα στα πλαίσια του διορθωτικού, της διορθωτικής επιστολής υπαριθμών 5. Ορισμένες διορθώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες επί της ουσίας, σαν παράδειγμα. Μπορεί να κάνει δημοσιονομικές προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017 σε σχέση με το 2016. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί επίσης και η διαδικασία επικύρωσης, αλλά αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. Τέλος, καλούμεθα να υιοθετήσουμε τους προϋπολογισμούς του συμπληρωματικούς 4 ε, και 5. Εμείς, το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο όμως ακόμα. Πάντως όλα είναι στη διάθεσή του έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει και στην αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και ο διορθωτικός προϋπολογισμός δείχνει ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Εξαρτώμεθα πολύ από τις επιθυμίες του Συμβουλίου έτσι ώστε ο προϋπολογισμός αυτός να γίνει δεκτός. Εξαρτώμεθα επαναλαμβάνω από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε στην διαπραγμάτευση. Απαιτείται να υπάρξει μια ταχύτατη διαδικασία και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδείξει διαθεσιμότητα, καλή πίστη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ταχύτατα μαζί του τον πολιετές. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Κύριε Καλβίνιο, παρακαλώ. Νομίζω μπορείτε να έχετε να απαντάτε στις, στα θέματα που έθεσε ο Γενικός Συγητής μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επισέλθω Στι λεπτομέρειε του σχεδίου διορθωτικού προβολισμού υπαριθμών 5 που έχει δύο πτυχε Το ένα αφορά τι συνολικέ μεταφορέ που γίνονται τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Είναι για πληρωμέ που δεν θα υλοποιηθούν. Άρα χρησιμοποιούνται εκεί που υπάρχει ανάγκη και δεύτερον έχουμε ενισχύσει κάποια προγράμματα α πούμε στο τμήμα 1α, στο 3 μέσω παραχρησιμοποίηση, μεταφορά λοιπόν κονδυλίων, ε, πιστώσεων από κεφάλαια του προπολισμού που δεν θα χρειαστούν. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά, δεν θα επισέλθω στι σχετικέ λεπτομέρειε, τα ξέρετε το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο αφορά τη μείωση, τη συνολική μείωση του προπολισμού λόγω τη καθυστέρηση, κυρίω τη καθυστέρηση ε, στην υλοποίηση του τμήματος 1β διαρθρωτικά ταμεία. Και εκεί ακριβώς κ. Φερνάντε έθεσε ερωτήματα. Τι γίνεται λοιπόν με τη μείωση κατά 7,3 δισεκατομμύρια του συνολικού προπολογισμού. Και δι, λόγω των μειώσεων, όπω είπα, στο τμήμα 1β. Έχουμε και μικρομειώσει από εδώ και από εκεί, όμω ακούστηκαν σχόλια για την γραφειοκρατία και ούτω καθεξής. Εγώ θα ήθελα, προκειμένου να καταθέσω τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Πρώτον, ας μην έχουμε αυταπάτες. Η αλλαγή από το N 1 στο N 3 άλλαξε την ταχύτητα υλοποίησης των διαθερικών προγραμμάτων. Χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία, περισσότερη ταχύτητα και αυτό ας μην το παραγνωρίζουμε. Όσον αφορά παραλαμβάνω το ρυθμό υλοποίησης που θα χαρακτηρίσει όλο το πι δελταπί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στο τέλος του αλλά και μετά το τέλος του. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Επίσης υπάρχουν εκ των προτέρων προϋποθέσεις μακροοικονομικές στο πλαίσιο του π.Δ.Π. δελταπί, τις γνωρίζει το Σκηνοβούλιο και υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις προαπαιτούμενα όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών δημιουργίας ε, θεσμών και μηχανισμών πριν πάρουν τα κονδύλια και αρχίζουν να τα Αυτό έχει επηρεάσει την ταχύτητα υλοποίηση. Είχε ω αποτέλεσμα κάποιε καθυστερήσει. Δηλαδή, τα προαπαιτούμενα είναι προαπαιτούμενα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουν ικανοποιήσει τι υποχρεώσει του τα κρατημέλη. Σημαντική προσπάθεια, απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα κρατημέλη. μην το υποτιμούμε αυτό. Και αυτό, επαναλαμβάνω, καθυστερεί την υλοποίηση του ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Ύστερα είχαμε καθυστερήσει στι εγκρίσει το είπε ο κύριος ε, Φερνάνδης, άλλους παράγοντες. Τέταρτον, διάφορα κράτη-μέλη. Ασχολούνται ακόμα με το κλείσιμο του 7-13 Τα υποστηρίζουμε όσο μπορούμε στην Κομισιόν για να αυξηθεί το ποσοστό πρόφησης για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 7-13. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο μέρος του... των προσπαθειών μας στοχεύει εκεί. Και τέλος, όντως ναι, παραδέχουμε ότι υπάρχει η ανάγκη απλούστευσης των κανόνων και συναφώς εμείς έχουμε καταθέσει φιλόδοξες προτάσεις, 15 νομοθετικά κείμενα και ο Σαρτουή αναφέρθηκε στην προσπάθεια αυτή. Άρα αυτή είναι μία πλευρά της εξίσωσης. Αλλά δεν θέλω να υπεραπλουστεύσω, δεν λέω ότι αυτή είναι μόνο οι λόγοι, μόνο οι λόγοι τους οποίους δεν υλοποιήθηκαν τα προγράμματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση Λόγω αυτών των καθυστερήσεων μειώνονται οι ανάγκε πιστώσεων πληρωμών στα διορθωτικά ταμεία. Σύμφωνοι. Εδώ προτείνουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις ανελήψεις υποχρεώσεων. Ε, μιλώ πάντα για το τροποποιητικό, τον διορθωτικό 4, έτσι. Λοιπόν, δεν λέω ότι οι αυξήσει αυτέ σε αναλήψει υποχρεώσεων είναι στο 7,3 δισεκατομμυρίων, αλλά στο τμήμα 3 τουλάχιστον για τους πρόσφυγες, την κρίση ασφάλειας και το προσφυγικό εκεί ενισχύουμε τις ε, πιστώσεις, ενισχύουμε κατά 15 και 10 εκατομμύρια αντίστοιχα πληρωμές και υποχρεώσεις. Ο κ. Φερνάνδες μάλιστα έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα προκειμένου. Αυτά τα 10 εκατομμύρια αρκούν. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση σας κύριε Φερνάνδες. Πιστεύουμε ότι επαρκούν. Στόχος αυτής της μικρής αύξησης είναι να προετοιμάσουμε για το χειμώνα τις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Πιστεύω ότι αρκούν τα 10. Αν χρειαστούν βέβαια περισσότερα θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Αλλά γι' αυτό προτείναμε τα συγκεκριμένα 10 και 15 εκατομμύρια. Επίση, όσον αφορά το Ταμείο του Ασύλου, και εκεί έχουμε προβλέψει αυξήσει. Ο Σιλβάνο θα σας πει περισσότερα αν χρειαστεί όσον αφορά τις δαπάνες για το, μείο, για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε λίγο πολύ προβλέψιμες ανάγκες. Και έχουμε κρεμεί αιτήματα από την Βουλγαρία, για παράδειγμα. Έχουμε επίσης τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω μετεγκατάστασης, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε προηγουμένω. Στο πλαίσιο του προπλογισμού του 2016, το μέσο ευελιξίας το έχουμε κινητοποιήσει πλήρω. και έχουμε και το περιθώριο πρόληπτες ανάγκες, το οποίο και αυτό κινητοποιούμε και θα κάνουμε το ίδιο και για το 2017. Βλέπετε προβλέπουμε και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Φερνάντες, Επίσης είπατε για τον εμπροστοβαρή χαρακτήρα του ΕΤΣΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό το ο χαρακτήρα χαρακτήρας δεν προδικάζει ουδόλω την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το έτσι για, το επόμενο, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το επόμενο πδπ Ήδη κάποιοι πόροι μεταφέρθηκαν στο 16 στο πλαίσιο του εμπροστοβαρούς αν θέλετε. Όμως να τονίσω για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση που έχουμε καταθέσει για το ΕΤΣΕΝ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το οποίο θα διαπραγματευτούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που ήθελα να καταθέσω. Να πω επίσης ότι υπάρχει πρόταση για την ενίσχυση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της Frontex. Εκεί προσπαθούμε να αυξήσουμε το προσωπικό, αλλά και αυτό δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες, αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Άκουσα και κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τα έσοδα. Έχουμε και εκεί μικροπροσαρμογές τον διορθωτικό 4, αλλά τα περισσότερα αφορούν τον διορθωτικό 5, γιατί εκεί έχουμε θέματα ιδιών πόρων. Να διευκρινίσω επίση ότι η διαδικασία κύρωση έχει ολοκληρωθεί. Η Ρουμανία ήταν τελευταία. Μα ε, ενημέρωσε τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωση από τα κρατημέλη. Η απόφαση για του ιδίου πόρου τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου. Με αυτά τελειώσαμε. Τώρα, χρειάζεται η αναπροσαρμογή των εσόδων στα κράτη-μέλη, σε διάφορα κράτη-μέλη. Όπω γνωρίζετε, η νέα απόφαση για του ιδίου πόρου θα ενσωματώσει το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσίων Λογαριασμών, το ΕΖΑ 2010. Υπάρχει μια μικρή μείωση του κόστου ίσπραξη παραδοσιακών ιδίων πόρων, όπω η δεσμοί προκειμένου. Και σιγά σιγά δρομολογούνται κάποιε επιστροφέ το είπατε αυτό, είναι κομμάτι της πολυπλοκότητας του συστήματος. Ευτυχώς εδώ έχω τον κύριο Λένερ και τον, Σέφερ, τον κύριο Σέφερ, οι οποίοι είναι ειδικοί επί του θέματος και θα απαντήσουν να χρειαστεί ερωτήσεις. Για να ληφθούν αυτά υπόψη λοιπόν, προτείνουμε το σχέδιο διευθυντικού προβολισμού 5. Ενημερώθηκατε τα μελη βεβαίω ναι, ήδη από την πρώτη αξιολόγηση επιπτώσεων τον Ιούλιο και τώρα του στέλνουμε πιο λεπτομερεί πληροφορίε αν έχουν προβεί σε προβλέψεις ε, για φέτος στο προπολισμό τους. δεν ξέρω ναι, τα κράτη-μέλη μας είπαν ότι ήδη έχουν προχωρήσει. Ίσως κάτι που δεν είχαν προβλέψει είναι οι μειώσει σε πληρωμές στο πλαίσιο του διορθωτικού 4. Αυτό προέκυψε όντω τις τελευταίες εβδομάδες. Όμως ε, για την απόφαση του ίδιου πόρου αυτά τα ήξεραν από την αρχή. Εάν ο διορθωτικός αυτός εγκριθεί φέτος, οι εθνικοί λογαριασμοί θα λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις για φέτος, όμως όσον αφορά τις πληρωμές, αν θέλετε τις χρηματοδομικές ροές, οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητέ ε, μάλλον τον Ιανουάριο και όχι τον Νοέμβριο. Εάν πάρουμε λοιπόν την απόφασή μας στην ε, Ολομέλεια του Νοεμβρίου, όπως είπατε, το συνολικό ποσό δεν αυξάνει, ότι παραπάνω εξοδεύσουμε πρέπει να το κόψουμε από κάπου αλλού. Αλλά αυτό, όπως είπα, για του εθνικούς λογαριασμούς θα φανούν τον Ιανουάριο. Θα ενσωματωθούν όμως στους εθνικούς προπολογισμού του 16 από πλευρά προπολογισμού, όχι cash flow. Κατά τα άλλα, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εγκρίνει τη σχετική απόφαση και τους δύο αυτούς για τα δύο αυτά σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καλβίνιο. Αν κατάλαβα καλά, ο συνάδελφό σα θέλει να πει δύο πράγματα για το Ταμείο για το Άσυλο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω την κατάσταση σχετικά με το Ταμείο Ασύλου ε, μεταναστεύσεως κλπ. Το ΑΖΙΦ δηλαδή, θα γυρίσω στα αγγλικά τώρα. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να υπενθυμίσω ότι το ΑΜΙΦ έχει τρία σκέλη. Αφενός οι χώρες μέλη και τα εθνικά προγράμματα, υπάρχει η επίγουσα βοήθεια και η δράση της Ένωσης. Αυτή η Emergency Assistance, το δεύτερο σκελός που χρησιμοποιείται για την ανταπόκριση σε ειδικές ανάγκες μέσα στη διάρκεια του έτους, εγγράφηκε στον προπολογισμό του 2016 με ένα ποσό περίπου 326 εκατομμυρίων, τα οποία απορροφήθηκαν όλα. Το ίδιο ισχύει και για τις δράσεις της Ένωσης, 43 εκατομμύρια για το 2016, τα οποία επίσης απορροφήθηκαν όλα. Το τι μένει τώρα ήταν στο πρόγραμμα για το ΑΜΙΦ, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την νομική του βάση, στα οποία ένα ποσό ενός δισεκατομμυρίου, 400 εκατομμυρίων σε υποχρεώσεις είχε εγγραφεί ήδη για το 2016 για να εφαρμοστεί με αποφάσεις του Συμβουλίου για τις μετεγκαταστάσεις, οι οποίες προέβλεπαν 160.000 προσώπων, μέχρι 160.000 δηλαδή προσώπων, τα οποία θα μετεγκαθίσταντο από την Ελλάδα στην Ιταλία. 640 εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί και διατεθεί στις χώρες μέλη για την μετεγκατάσταση στα πλαίσια στη διάρκεια δηλαδή του έτους περίπου 200 εκατομμύρια που παρέμεναν διαθέσιμα στις υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν στο νέο εργαλείο στήριξης εσωτερικής ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό ε, προσφύγων που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου 2016, ενέκρινε το Συμβούλιο απόφαση για να επιτρέψει στις χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των χρημάτων που προβλέπονταν για τις μετεγκαταστάσεις για την χρηματοδότηση του προγράμματος που είχε συμφωνηθεί με την Τουρκία, στη συμφωνία δηλαδή μέσα με την Τουρκία, που επιτρέπει την επανεγκατάσταση προσώπων που επιστρέφουν στην Τουρκία και πρόκειται να επανεγκατασταθεί σε χώρα μέλος. Η απόφαση αυτή καλύπτει μέχρι 54.000 άτομα τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν, με εγκατασταθούν να μάλλον από την Τουρκία σε χώρες μέλη. Ένα μέρος των χρημάτων που προβλέπονταν αρχικά για τις μετεγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αυτή την έναν προς έναν επανεγκατάσταση σε χώρα μέλος. Αυτά που μένουν τώρα είναι μια υπόμνηση των αρχικών κονδυλίων για το ΑΜΥΦ είναι 200 περίπου εκατομμύρια, τα οποία θα αναμένεται να απορροφηθούν πλήρως μέχρι τέλους του έτους και θα χρησιμοποιηθούν για επίγουσα βοήθεια, emergency assistance, που αυτή τη στιγμή βασίζεται σε αιτήσει των χωρών μελών και έχει ζητήσει στον διορθωτικό προϋπολογισμό 4 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση του ΑΜΙΦ κατά 130 εκατομμύρια στις υποχρώσεις. Χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση άλλων αναγκών ενδεχομένως μέχρι τέλους του έτους. Σε μια κατάσταση μέσα που παραμένει αρκετά ασταθής σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές και τους ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στα νότια σύνορά της. Με τα λόγια αυτά και με τις αυξήσεις που έχουν ζητηθεί για το στον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 4, πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες είτε γνωστές είτε αναμενόμενες μέχρι τέλους του έτους 2016. Σας ευχαριστώ κύριε εσείς κύριε Φερνάντες. Απαντήθηκε η ερώτηση σας εσείς κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνολικά συμφωνώ με τα ερωτήματα του Φερνάντες. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές είχα πει κάποια στιγμή ότι αρνούμε να ασχοληθώ πλέον διότι Κάποτε ζητούμε παραπάνω χρήματα, τώρα εδώ μένουν αδιάθετα 7 δισεκατομμύρια. Όποιο και αν είναι ο λόγο. Είτε πρόκειται για καθυστέρηση από πλευρά χωρών μελών, είτε πρόκειται για ε, διοικητικέ παραλήψει και τα λοιπά, είναι πολύ αρνητικό για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό, ένα πραγματικό πρόβλημα και καλώς κάνουμε και προβλέπουμε ή θα προβλέψουμε μια ε, συνάντηση για να δούμε τι θα γίνει με, το, με τα χρήματα αυτά. Αυτό το γιογιό θα συνεχιστεί και περισσότερο ίσως διότι θα περάσουν μήνες και μέχρι τέλους της θητείας για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Τώρα για την κρίση του μεταναστευτικού που με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι προβλέπονται πρόσθετα κονδύλια ακούγοντα τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γεγονό ότι δεν μα κοστίζει παραπάνω είναι διότι κάποιε πολιτικέ δεν λειτουργούν. Διότι αν οι πιστώσει που είναι αναγκαίε για την επανεγκατάσταση δεν χρησιμοποιούνται, τα ποσά επίση για την μετεγκατάσταση δεν θα σα αναφέρω τι λεπτομέρειε των ποσών τώρα, διότι καθίσατε τελικώ και ακριβότερη κατάσταση από την επανεγκατάσταση. Όλα αυτά δημιουργούν βέβαια ένα περιθώριο, αλλά είναι λόγω τη αποτυχία των σχετικών πολιτικών. Και χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα. Και αυτό χρειάζεται κάποια μελέτη. Τέλος και χωρίς να θέλω να είμαι προκλητικός, όταν μιλούν για DAB 4, προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, και θυμίζουμε την κατάσταση της Μεγάλης Βρετανίας. Αν τα κατανοώ καλά, αποφάσισε η Μεγάλη Βρετανία να καταλήψει την Ένωση, υπάρχουν τώρα χώρες μέλη, οι οποίες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν έξτρα χρήματα για τον διορθωτικό μηχανισμό. Αν κατάλαβα καλά. Αν δεν κατάλαβα καλά, ζητώ συγγνώμη. Εκπλήσωμε από αυτά που προβλέπονται σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε αν κατάλαβα καλά ή όχι. Έχασε λοιπόν αξία η Βρετανική λίρα όταν, ε, όταν αποφασίστηκε η έξοδος. Οι Βρετανοί αποφάσισαν να εξέλθουν, αποφάσισαν ε, να προχωρήσουν στο Brexit. Και θα χρησιμοποιηθεί τώρα το προϊόν των προστήμων για να αντισταθμίσουν την απώλεια της ε, Βρετανικής λίρας, αξίας Βρετανικής Λύρας δηλαδή, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα κληθούν οι χώρες μέλη να το πληρώσουν αυτό, να μου το εξηγήσουν αυτό. Όταν λένε οι Βρετανοί φεύγουμε, χάνει 20-30% αξία, άρα μειώνεται και η αξία της Βρετανικής συμβολής και τι λένε, α όχι δεν είναι Βρετανικό πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα των υπολείπων. Μα, τι να πω. Διερωτώ με λοιπόν. Υπάρχει πάντως και κάτι θετικό μέσα σε όλο αυτό το μηχανισμό των προστήμων, ότι δηλαδή πάντοτε ζητούσαμε εμείς το προϊόν των προστήμων να παραμένει μέσα στον προϋπολογισμό και να μην επιστρέφεται στις χώρες μέλη. Αλλά ε, κοιτάξτε, εδώ είναι εκπληκτικό αυτό που προτείνεται. Ή μήπω κάνω λάθος και δεν έχω κατανοήσει καλά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξεταστεί η υπόθεση αυτή και πάντως με μεγάλη πρόσοχη. Πρόεδρος, μπορούμε να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τι γίνεται με τη Μεγάλη Βρετανία. Θυμούμε τον Φεβρουάριο όπου ο τότε Πρωθυπουργός Κάμερον έλεγε Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε η Ευρώπη να έχει μονάχα ένα νόμισμα. Εμεί ζητούμε και επιμένουμε να υπάρχουν πλέον νομίσματα. Όταν λοιπόν ρυθμίζεται η συνεισφορά τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία καταβάλει τη συνεισφορά τη σε λίρε, στερλίνε, υποθέτω ότι υπάρχει κάποια ισοτιμία μεταξύ στερλίνα και ευρώ. Πότε ε, καθορίζεται αυτή η ισοτιμία και τι γίνεται στην περίπτωση, διότι αν κατάλαβα καλά, θα υπάρχει την στιγμή της πληρωμής ένα έλλειμμα 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Άρα την ζημία την υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα το 2016 όπου το Brexit ήδη κακοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς το εξηγείτε αυτό. Διότι κανονικά η Μεγάλη Βρετανία θα έπρεπε να πληρώνει σε ευρώ Κάποια στιγμή όμως είχε καθοριστεί κάποια ισοτιμία. Μπορεί να διευκρινίσει κάπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να περιμένουμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Ντουνανού. Πρόκειται για ένα πραγματικό ερώτημα ουσίας. Εγώ πάντως θέλω να παρέμβω πρώτα για να πω στον κύριο Φερνάντες ότι χρειάζεται καλείται να είναι πιο ευανάγνωστο για τον ε, ε, Ευρωπαίο πολίτη. Ο προπολογισμό τη Ένωση είναι αφόρητο να μην μπορεί κανεί να κατανοήσει τι σημαίνει ο προπολογισμό του σύνολό του. Επανέρχομαι ωστόσο σε αυτή την απόκληση μεταξύ ε, υποχρεώσεων και πληρωμών. Και κάθε χρονιά βλέπουμε το ίδιο. Γνωρίζω και από εμπειρία, επειδή έχω ασχοληθεί με τα διαφορετικά ταμεία πολύ καιρό, ότι χρειάζονται δύο χρόνια ανάμεσα στην αίτηση και στην καταβολή του ποσού από την Ευρώπη. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Είναι υπερβολικά περίπλοκα τα κυκλώματα και αυτές οι καθυστερήσεις ε, αποθαρρύνουν τον κόσμο που τον Και μια ερώτηση για την αιρεσιμότητα. Εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου όπου λέει ότι η Ισπανία και Πορτογαλία δεν σέβονται τους όρους της μακροοικονομικής ερεσιμότητας και για το λόγο αυτό αναστέλλονται τα διαφθορτικά ταμεία. Εκπλήσωμαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν επελήφθη του θέματος. Είναι παράξενο. οι ε, Ρεζή και Κοντ να ασχολούνται με το θέμα αυτό, ενώ είναι προφανής ή δημοσιονομικές επιπτώσεις από το θέμα αυτό. Επιθυμώ να μάθω λοιπόν για ποιο λόγο η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν συμμετέχει στην απάντηση που δίνεται στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος Αρτουή. Η επιστολή που έστειλα στον πρόεδρο είχε ως αντικείμενο να, να πούμε ότι έδειξαν μια υπερβολική επίκη απέναντι στην Ελλάδα και γιατί άραγε είναι διαφορετική μεταχείριση της Ελλάδος από αυτήν της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Κύριε Ντεπρέ, πρόσθετο σχόλιο. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα χρειαστεί να καταβληθούν για την αντιμετώπιση της απώλειας της αξίας της λίρας τερλίνας πρέπει να αφαιρεθούν 9 εκατομμύρια διότι σε άλλο σημείο του εγγράφου, το DAB 4 λέει ότι επειδή η European Medicine Agency που είναι εγκατεστημένη στο Λονδίνο θα χρειαστεί σε αυτήν να πληρωθούν 9 εκατομμύρια λιγότερα. Ας μου εξηγήσουν και αυτό. Κοιτάξτε, πρέπει ναι, να διατηρήσουμε όλα τα όλους, όλα τα, όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί λόγω χάρη μάλλον στην ε, υποτίμηση της Λίδας, θα μας κοστίζουν και λιγότερο. Έτσι δεν είναι κύριε Χουντή. Πρόεδρος, Κομισιόν, παρακαλώ. Σε ποια χρονική στιγμή καθορίζεται η ισοτιμία στερλίνας ευρώ. Γιατί αν είχε ανέβει η στελίνα θα ήμασταν... Είχαμε και κάποιο κέρδος. Κύριος Φερνάντες, επιπλέον ερώτηση. Δεν υπάρχει υποτίμηση της στελίνας; το καρτιμέλι πλέον περισσότερο. Εάν ανέβει η Στερλίνα σε σχέση με το ευρώ, αυτά τα χρήματα που ενδεχομένω κερδίζουμε επιστρέφουν στον προπολίσμο ή υπάρχει ανώτατο όριο, δεν, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή η ανατίμηση. Πρόεδρος. Όπως είπα, είμαστε σχεδόν ανίκανοι να διαχειριστούμε αυτόν τον προπολισμό έτσι όπως είναι. Κομισιόν, Πρόεδρε. Είναι χαρακτηριστικό των εσόδων του προπολισμού, του ευρωπαϊκού προπολισμού. Οι συνεισφορές των κρατών μελών είναι καθορισμένες, καθορίζονται μάλλον στο τέλος του ημερολογιακού έτους, όταν ψηφίζεται ο προπολισμός από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κανονικά 31 Δεκεμβρίου έτους του προηγουμένου έτους, δηλαδή από το έτος του προπολογισμού. Συνεπώς, οι ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συνεισφορών των κρατών μελών που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ είναι ισοτιμίες που της 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Δηλαδή για το 16 καθορίστηκαν είναι οι ισοτιμίες αν θέλετε της 31ης Δεκεμβρίου του 2015. Εν τούτες, οι πραγματικές συνεισφορές δεν γίνονται άπαξ στην αρχή του έτους αλλά κατά 12 τιμόρια ένα, ή κατά ένα ή δύο 12 κατημόρια, εν πάση περιπτώσει ε, εκταμιεύονται κατά τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς, μπορεί να προκύψουν διαφορές λόγω της διαφοράς της ε, συναλλαγματικής οτιμίας που χρησιμοποιήθηκε για προϋπολογισμό και την πραγματική αξία των συνεισφορών όταν εισπράττονται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτές οι διαφορές φυσικά ε, μπορεί να είναι προ τα πάνω προ τα κάτω. Το 2015, κατά τη διάρκεια του 2015, η Στελίνα είχε ανέβει. Είχε ανατιμηθεί Συνεπώ, στο τέλο του έτου, και δεν θυμάμαι το ακριβέ πόσο, είχαμε κάποιε εκατοντάδε εκατομμύρια. Τα έχουμε κερδίσει σε ευρώ, χάρη στη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στι από Ανάποδα γίνανε τα πράγματα το 2016. Η Στελίνα υποτιμήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016. έχουμε, έχουμε μεγαλύτερη υποτίμηση, πτώση της τιμίας όσο περνάει ο χρόνος και θεωρούμε ότι θα έχουμε μια αρνητική διαφορά στο τέλος του έτους, δηλαδή σε ευρώ αν θέλετε θα έχουμε σπλάξει λιγότερα ευρώ από ό,τι είχαμε προβλέψει, θα έχουμε καθαρή απώλεια. Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής. Κέρδη οι ζημίες αφορούν το κράτος μέλος. Δηλαδή το κράτος μέλος πλέον περισσότερα ή λιγότερα. Αν υπάρχουν ε, απόλυτε βεβαίω, υπάρχει κίνδυνο στο τέλο του έτου, στο κλείσιμο αν θέλετε, να έχουμε έλλειμμα όσον αφορά τον προπολισμό και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Συνεπώ, κρατούμε κάποια ποσά από πρόστιμα για να αντισταθμίσουμε την αναμενόμενη απώλεια εσόδων σε ευρώ. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφής. μία διευκρίνηση. Γιατί δεν βάζετε στις τροποποιήσεις που παρουσιάζετε τα πραγματικά ποσά των έκτακτων εσόδων που είναι τα πρόστιμα και το 1,8 δις από την υποτίμηση της Τερλίνας. Γιατί εσείς προχωράτε στην αντιστάθμιση των ποσών. οι συνεισφορές οι δημοσιονομικές ανταποκρίνονται σε δαπάνες τελικά. Καλύπτουν δαπάνες. Αν υπάρχει μια απώλεια από τη συναλλαγματική ισοτιμία τέτοιου είδους που θα σημαίνει ότι δεν καλύπτονται όλες οι δαπάνες από έσοδα, τότε στο τέλος θα είχαμε ε, στα πλαίσια του κλεισίματος του προϋπολογισμού ένα έλλειμμα και νομίζω ότι μέχρι τώρα πάντα είχαμε πλεονάσματα. Αν όμως φτάσουμε σε αυτή την ακραία κατάσταση και έχουμε έλλειμμα, τότε το έλλειμμα θα πρέπει να καλυφθεί από νέες συνεισφορές τον επόμενο χρόνο. Αυτό θα είναι δυσάρεστη κατάσταση γιατί θα μειώσει επιστώσεις πληρωμών για το 17. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς να έχουμε μια ισορροπία για το 16 σε επίπεδο εσόδων, πόρων και νομίζω ότι ένα τμήμα των προστήμων θα χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Να προσθέσω εδώ ότι αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε είναι να υπάρχει μια ρύθμιση προς μια κατεύθυνση η οποία στο τέλος θα πρέπει να αντιστραφεί. Λοιπόν, σε σχέση με τον υπολογισμό των, του ΑΕΠ της ε, κάθε χώρας, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μία πορεία βασισμένη πάνω στα ΑΕΠ των χωρών και στο τέλος να αναγκαστούμε να πάμε ανάποδα, να κάνουμε το αντίθετο. Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι η διαφάνεια. Ε, σε επίπεδο πόρων έχουμε να κάνουμε με, αν θέλετε, με ένα καλάφι στο οποίο μπαίνουν και τα κράτη-μέλη, υπάρχει ένα περίπλοκο συμβούλιο, κάποιες χώρες προσπαθούν να πάρουν επιστροφές. Αν η συζήτηση αυτή γινόταν δημόσια, δεν θα υπήρχαν τέτοιου είδους μικρορυθμίσεις ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνεται σε δημόσιο επίπεδο. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατικό. Σαν να λέμε δεν είναι δική σας υπόθεση, είναι υπόθεση των 27 χωρών. Επιβεβαιώστε μου λοιπόν. Δεν μπορώ να δώσω εγώ αυτή τη στιγμή την ικανότητα να απαντήσω, αλλά στην διορθωτική 4 λέτε εσείς ποιο είναι το πραγματικό ποσό το οποίο είναι προϊόν προστήμων και ξεπερνάτε το 1,8 για την πιθανή υποτίμηση της τερλίνας. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ότι ήταν ιδιαιτέρως ε, διαφανές. Στην διορθωτική 4 δεν το κάνουμε, δεν προτείνουμε να το κάνουμε. Λέμε ότι εμείς δεν θα δημοσιονοποιήσουμε τις, ε, δεν θα εντάξουμε στον προϋπολογισμό τα πρόστιμα αν τα χρειαστούμε Συνεπώς λοιπόν τα πρόστιμα δεν περιλαμβάνονται στο 4, μα αυτό δεν είναι κανονικό. Τα βάζετε στην άκρη. Θα πρέπει να υπάρξει και ένας ε, ε, συμπληρωματικός 6 όταν έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία σαν παράδειγμα από την πραγματική υποτίμηση της Τερλίνας. Κοιτάξτε, τα υπόλοιπα δεν θα έρθουν μέσα από ένα διορθωτικό προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα είναι ακριβώς αυτό το πλεόνασμα ή το έλλειμμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Λέναρντ. Κάθε χρόνο, τον Απρίλιο περίπου του επόμενου χρόνου, δημοσιεύουμε το τελικό αποτέλεσμα των ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ελλείμματα και δεν θέλουμε να έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε υπερβολικά διαφανείς. Λέμε ότι υπάρχουν κάποια πρόστιμα, έχουν πραγματικά τελεσικήσει, αλλά εμείς δεν τα εντάσσουμε γιατί τότε θα είχαμε ε, πιθανότητα αύξησης ενός ελλείμματος, κάτι το οποίο θα θέλαμε να αποφύγουμε. Ο κύριος Δεπέ. Κοιτάξτε, εγώ Είχα κάνει μια παρατήρηση παράλογη, αν θέλετε, σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή μια χώρα θέλει να φύγει και τότε οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιβαρυνθούν για τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην εξοδότηση. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν των προστήμων μένει στον προϋπολογισμό αν καταλαβαίνω καλά θα το αφήσει στον προϋπολογισμό σαν αντιστάθμιση ε, της ηλικιότητας ε, την οποία θα κάνουμε αντισταθμίζοντας το κόστος της Βρετανικής εξόδου. Κοιτάξτε όπως και να έχουν τα πράγματα. Εάν τα πρόστιμα φανούν ως έσοδα, τότε θα τα έπαιρναν απευθείας ε, τα κράτη-μέλη στον προϋπολογισμό τους και στο τέλος του χρόνου θα είχαμε πράγματι ένα έλλειμμα. Οπότε θα έπρεπε να ζητήσουμε από τα κρατη να μας τα δώσουν πίσω για να αντισταθμίσουμε το έλλειμμα. Νομίζω ότι θα ήταν σωστότερο να πούμε ότι η ζημία σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία είναι ε, το κόστος της εξόδου. Ήδη το κόστος έχει φτάσει το 1 δις 800 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Είναι σαφές αυτό. Ενθυμίστε, ενθυμίστε ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου είχε δεκτεί τον Φεβρουάριο ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα υπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ρίξει κάποιο φως. Ο κύριος Γκάιερ έχει στήσει το λόγο. Ένα σχόλιο που δεν το εννοώ και απόλυτα σοβαρά. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα στην εφημερίδα Financial Times, αλλά είδα και, μάλλον, μάλλον με είδαν και χθε δημοσιογράφοι και με ρώτησαν αν όντω η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται σοβαρά 42.000 μπουκάλια κρασί, τα οποία βρίσκονται φαίνεται σε κάποιο υπόγειο είτε της Κομισιόν είτε του ε, Συμβουλίου, αν πρόκειται να ζητήσει το μεριδιό τη η Μεγάλη Βρετανία από αυτά τα 42.000 μπουκάλια κρασί. Έχω μια πρόταση. Μπορούμε τότε να πάμε κι εμείς στην Βρετανική μόνιμη αντιπροσωπεία και αν μας κάνει τόσες δυσκολίες με αυτό το Brexit η Μεγάλη Βρετανία να ζητήσουμε κάποια τι μορφή. Ε, δηλαδή κάποια αποζημίωση είδος από την ε, ε, κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητας. Να πάμε δηλαδή να κολλήσουμε σημεούλες Ευρωπαϊκής Ένωσης απάνω στα αντικείμενα αυτά για να πούμε ότι να, με αυτόν τον τρόπο θα ισοφαρίσουμε κάποιες από τις ζημίες που υφιστάμεθα από την έξοδό σας. Αυτή είναι η δική μου ιδέα. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ. Qui fait partie du patrimoine quand il y a Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο θα πρέπει να υπάρξει διαμοιρασμός της περιουσίας. Και δεν νομίζω ότι οι Βρετανοί θα πάρουν μέρος στην ανακαίνιση του συγκεκριμένου Βελγικού Μουσείου. Και φυσικά ούτε καν στην λειτουργία του συγκεκριμένου Βελγικού Μουσείου. Καλό. Λοιπόν, κύριε Φερνάντες, για Συμπεράσματα. Συμπεράσματα μπορούμε εμείς να καταστήσουμε όμοιρο το διορθωτικό 4 στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το ε, πολιετές δημοσιονομικό και για τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό του 17. Το Συμβουλίο ζήτησε να ψηφίσουμε τον ΤΑΠ 4, τον συμπληρωματικό 4, τον Οκτώβριο 2 στο Στρασβούργο. Ίσως θα μπορούσαμε εμείς να ζητήσουμε η διαπραγμάτευση να γίνει από κοινού DAB 4, DAB 5, διορθωτική δηλαδή 4 και 5, εγγύηση για τους νέους και επίσης προϋπολογισμός του 17. Τότε σε αυτή την περίπτωση, λέει ο κύριος Φερνάντες, θα πρέπει να περιμένουμε τη θέση του Συμβουλίου, την οποία δεν γνωρίζουμε. Εμείς είμαστε γεμάτοι καλή πίστη, γεμάτοι καλή θέληση, είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε την μπάλα την έχει το Συμβούλιο. Αν το Συμβούλιο πραγματικά θέλει να παίξει παιχνίδι, τότε είμαστε έτοιμοι. Αν το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, αλλά αυτοί πρέπει να μας πούνε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Και φυσικά όλα τα θέματα εδώ συνδέονται μεταξύ τους, όπως ακριβώς είπατε. Και όταν ένας Πορτογάλος μιλάει για ποδόσφαιρο, για μπάλα, φυσικά κάτι ξέρει. Είναι έτοιμος να σκοράρει, αστείευεται ο πρόεδρος. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουλίν για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε έτσι ώστε να δοθεί επίγουσα βοήθεια σε περίπτωση εθνικών καταστροφών. Ο κανονισμός όπως τροπολογήθηκε το 2014 δίνει την δυνατότητα μέχρι 50 εκατομμύρια να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό σε επίπεδο πιστώσεων πληρωμών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των ποσών αυτών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Το Ταμείο αυτό δεν είναι μόνο οικονομική βοήθεια, είναι σαφές πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης στους πολίτες που έχουν φυγεί. Επιτρέπει να δοθεί η βοήθεια αυτή το ταχύτερο δυνατόν η ικανότητα άμεσης απόκρισης θα δώσει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει την βελτίωση της παρέμβασής της στο μέλλον και γι' αυτό ζητώ από όλους να στηρίξετε την πρόταση για την ένταξη του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και τη σύσταση. Θέλει κανείς το λόγο. Όχι, από φαίνεται. Τροπολογίες για την έκθεση κυρία Σουλήν. πρέπει να κατερθούν πριν από τις 10 το πρωί της 14 η Οκτωβρίου. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει 9 ή 10 Νοεμβρίου και δεν ξέρω πότε θα πάει στην Ολομέλεια η έκθεση. αλλά σίγουρα εντός του 16. Λόγος στον κύριο Βίκτορ Νεγκρέσκο να αφορά το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για μια υπόθεση στην Εσθονία. Η Petroleum and Chemicals. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. 11 Μαΐου του 2016 η Εστονία επέβαλε αίτηση για συνδρομή από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση για πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Σχετικά με 1550 εργαζομένους που απολύθηκαν. 800 εξ αυτών ε, είναι δυναμή δικαιούχη. Η Εστονία, η οικονομία της Εστονίας ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι εξαγωγές και οι απολύσει αυτέ έγιναν σε μια περιοχή στα βορειοανατολικά της ε, Εστονία που υπέφερε τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια λόγω της αναταραχή στην αγορά πετρελαίου. Λόγω επίση της μεγάλη απόστασης ε, από το κέντρο. Η έκθεση Επίσης, αναφέρεται στην παραγωγή χημικών προϊόντων στην Ευρώπη, η οποία μειώθηκε κατά πολύ σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό. Επλήγει λοιπόν ο τομέας. Η αίτηση βάλετε στα πλαίσια και με τήρηση των κανόνων του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση. Η αίτηση είναι συμβατή με όλους τους ε, κανόνες και τις προϋποθέσεις που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων για τον εφορικό χαρακτήρα της οικονομίας. Προτείνω λοιπόν α, ότι προτείνω θα καλούσα τους συνεδέλφους να απόσουν από προσθήκη πολιτικών σχολείων στην έκθεση που δεν υπηρετούν τον συγκεκριμένο στόχο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συστούμε ο κύριος Ταράν. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Χαίρομαι που ήλθε η έκθεση στο τραπέζι μας. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ναι, ε, δεν θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές πτυχές του Ταμείου. Καλό και εγώ τους συναδέλφους και την γραμματεία. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την έκθεση και να στείλουμε το σχετικό μήνυμα, να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν για ενεργά μέτρα στα αγορά εργασία και ότι δεν χρηματοδοτούν τον υπερπολισμό της Εστονίας. Όχι, πηγαίνουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους ανέργους που μπορεί να μην ξέρουν πώς λειτουργεί το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Ούτε προσπαθούμε να ξεπλύνουμε τις αμαρτίες, τις περιβαλλοντικές αμαρτίες μιας βιομηχανίας. Λοιπόν, ο Σάρφος Ούρμας και εγώ είχαμε μιλήσει στην ε, ιστορική κυβέρνηση και τους είχαμε ζητήσει να δώσουν χρήματα για το Ταμείο και μας είπαν όχι έχουμε αρκετά χρήματα από μόνοι μας και να που ένα χρόνο μετά έρχονται εδώ ζητώντας. Βλέπετε λοιπόν ότι η Επιτροπή μας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και να ασκήσει επιρροή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συγχαίρω όλους όσους ασχολήθηκαν με την Εστονία και Σπέιτ. Πρόεδρε, και εγώ προσθέτω ότι είναι η πρώτη φορά που η Εστονία ζητάει κάτι από το συγκεκριμένο ταμείο. Και εγώ προσωπικώς ε, το βλέπω σημαντική εξέλιξη. Δυστυχώς συνέβησαν πράγματα, συμβαίνουν, για τον τομέα των χημική της, στη, της χημικής βιομηχανίας στη συγκεκριμένη περιοχή της Εστονίας αλλά έτσι είναι η αγορά του πετρελαίου έτσι είναι οι τιμές αυτήν την αγορά έτσι είναι η βιομηχανία, η τεχνολογία και κάποιοι επηρεάζονται ευθέως από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια. Η περιοχή της Εστονίας από κοινωνικής απόψεως είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Γι' αυτό και η ενίσχυση από εμάς, από το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται για πρακτικούς αλλά και συμβολικούς, ψυχολογικούς θα έλεγα λόγους ως επίδειξη αλληλεγγύης. Και να τονίσω επίσης ότι εφόσον εγκρίνουμε το μέτρο, τα σχετικά ποσά θα διατεθούν για μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας. Πρώτος ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Το θέμα είναι το Ταμείο να μπορεί να παρεμβαίνει και δεν το λέω για να το υποτιμήσω ε, πριν ε, αντιμετωπίσουμε τέτοιες ενεργών και όχι μετά, όχι εκ των υστέρων. Κύριε Νεκρέσκου, έχετε κάτι άλλο να πείτε, όχι. Οπότε, η Επιτροπή Επασχόλησης θα ψηφίσει αύριο, 12 Οκτωβρίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 13 Οκτωβρίου Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει στις 14 και μετά πάμε βεβαίως στις 26 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια όπου θα τεθεί προς ψηφοφορία το κείμενο. Και τώρα... γιατί όσον αφορά τις ροές προσφύγων και μεταναστών αντιμετώπιση των μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Βιώτη. Όπως είπατε η γνωμοδότηση την οποία προετοιμάζουμε είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΔΕΒΕ και την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Η λεγόμενη μετασταθευτική κρίση, λέει ο μιλητής, δημιουργεί θέματα και όχι μόνο πολιτικούς, πολιτικής φύσεως, αλλά δείχνει μια έλλειψη πόρων και ευελιξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιετές πλαίσιο ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν καταστάσεις υψηλής δυσκολίας. Συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να βρουν λύσεις εκτός κοινοτικού προϋπολογισμού, λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές, γιατί σαν παράδειγμα το Ταμείο για την Αφρική είναι κάτι το θετικό. Η, η χρηματοδότηση των αναγκών των σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Το θέμα είναι βέβαια ότι τα ταμεία αυτά διαφεύγουν του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί είναι έξω από τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο βασικός στόχος των διαθεσίμων μέσων και γιατί ακριβώς εμείς θα πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μόνο των συνόρων όλων των χωρών προέλευσης. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ρίζα του. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την φτώχεια των περισσότερων αυτών χωρών και γι' αυτό ακριβώς τα βήματα που προτείνει για διάλογο με την Αφρική η Επιτροπή είναι θετικά και προσφέρει νομίζω δυνατότητες ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να σταματήσουμε τις πηγές της μετανάστευσης, πώς θα ειρηνεύσουμε τη Μέση Ανατολή και θα, πώς θα αναπτύξουμε την Αφρική. Η κυρία Γιάτεμα και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πράγματι ευαίσθητο και δύσκολο το θέμα. Δύσκολο για την Επιτροπή μας άλλωστε να ανταποκριθεί ε, σε τέτοια θέματα. Η χρηματοδότηση των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης είναι το αντικείμενο της εκθέσεως. Η δε διάθεση πολλών από τα κονδύλια αυτά κοίται εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εάν δαπανούμε χρήματα ωστόσο των Ευρωπαίων φορολογουμένων, κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Εάν δηλαδή δημιουργούνται ταμεία τα ταμεία αυτά θα πρέπει να υπάγονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο με κάποιο τρόπο. Εμείς δε θα πρέπει νομίζω να κρίνουμε και να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα ασκείται ο κοινοβουλευτικό έλεγχος. Ήσταμε κριτικά απέναντι σε τέτοια ταμεία. Ωστόσο, κατανοώ ότι υπάρχουν λόγοι που τα υπαγορεύουν, υπαγορεύουν τη δημιουργία τους, χρειάζονται κεφάλαια για την ε, Αφρική. Όμως χρειάζονται πιο ξεκάθαρες αιτιολογήσεις, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι και πότε. Εάν δηλαδή η δημιουργία και χρηματοδότηση μέσω ταμείων εξαρτάται από την καλή θέληση κάποιων, αυτό δεν μου αρκεί. Δεν αμφισβητώ την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αιτίε της μεταναστεύσεως, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσπάθεια αυτή με βρίσκει αντίθετη. Πρέπει να διασφαλίσουμε στις χώρες αυτές ανθρώπινα δικαιώματα και αηφόρο ανάπτυξη. Αυτά πρέπει να λυθούν οπωσδήποτε υπόψη. Η διαφάνεια και η απόδοση λογαριασμών είναι απαραίτητα. Οι αρχές αυτές είναι ουσιώδους σημασίας και πρέπει να ισχύουν και να γίνονται σεβαστές σε κάθε διάθεση κονδυλίων. Ευχαριστώ κύριε Γιάτριν Μάκη, λέει ο πρόεδρος Αρτουή. Ασφαλώς και μας ανησυχεί αυτή η ραδέα αύξηση του προϋπολογισμού αλλά και το γεγονός ότι δεν είναι εύληπτος για τον ε, πολίτη. Ο προϋπολογισμός δεν έχει και τα αναγκαία μέσα για να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες και επομένως εν μέρη διαφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν ζητεί άλλο τον λόγο. Εσείς κύριε Βιώτη επιθυμείτε να λάβετε και πάλι το λόγο όχι. Άρα, μένει να σας πω ότι στις 19 Οκτωβρίου, 10η πρωινή, μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε ε, τροπολογίες στο έγγραφο του κ. Βιώτη. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολισμών θα γίνει στις 9 ή 10 ενδεκάτου και θα διαβιβαστεί η έκθεση, σημαντική αυτή η έκθεση και που έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, στην Επιτροπή Εξωτερικών που συνδιασκέπτονται στην βάση του άρθρου 55 για ε, εξέταση και ελπίζω ότι θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους το περιεχόμενο της γνωμοδοτήσεώς μας. Η έκθεση της κυρίας Φενάντες η κυρία Γκουάρια Ζαμπάλ δηλώνει για τη σχηματοδοτική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρεί λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο και άλλωστε είμαστε συναρμόδιοι και με την Επιτροπή Οικονομικών. Άρα αναβάλλεται η έκθεση αυτή και έτσι λοιπόν εγώ θα διακόψω τις ε, δραστηριότητες μας οι οποίες θα επαναληφθούν από τις 3 το απόγευμα. Υπενθυμίζω ότι η περίοδος ψηφοφοριών αρχίζει στις 4 το απόγευμα. Διακόπτω τη συνεδρίαση.